Good afternoon, everybody. And you are most welcome to this. Uh, Καλό απόγευμα σε όλους. Καλώς ορίσατε στο εργαστήρι. Θα μιλήσω σχετικά τώρα. Αν τυχόν δεν καταλαβαίνετε σουηδικά, πάρτε και τα ακουστικά για να με καταλάβετε. μία τα Stark. <laughs> Okay, Ξανά λέω στα Σουηδικά. Καλώς ορίσατε. Ε, και συμβαίνει στο πλαίσιο διαφόρων δραστηριοτήτων ε, του Κοινοβουλίου. Ο στόχος είναι να συζητήσουμε το θέμα της ανεργίας εν γέννη. Στις 20 ε, Μαρτίου η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς ε, διοργάνωσε ένα σεμινάριο για διάφορους τρόπους εξόδου από το πρόβλημα. Η Επιτροπή Απασχόλησης συζήτησε ε, το ενδεχόμενο σύνταξη μιας νέας έκθεσης πρωτοβουλίας του Κοινοβουλίου για να συμμετάσχουν περισσότερο οι νέοι στην αγορά εργασίας ε, πολλές τέτοιες δραστηριότητες δεν ενσωματώνουν την διάσταση του φύλου ε, σε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες που προανέφερα και άλλες. Ε, παραγνωρίζεται γενικώ η σημασία αυτής της διάστασης στις πολιτικές συζητήσεις και γι' αυτό αποφασίσαμε να διοργανώσουμε το σημερινό σεμινάριο Χαιρόμαστε που η συγγήτριά μας, η κυρία Αντζελίλη, είναι μαζί μας σήμερα. Το εφαλτήριο ήταν η ανάγκη του να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας πόσο διαφορετική είναι η κατάσταση που βιώνουν οι γυναίκες και οι άντρες ε, αντίστοιχα και πώς πρέπει να προσαρμόσουμε την κατάσταση για να επιτύχουμε ε, τους ευρύτερους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μας μιλήσουν τα μέλη του πάνελ για τη διακριτική μεταχείριση, στην κατάρτιση, στην αγορά εργασία, στην πρόσβαση, στην κοινωνική ασφάλιση, γενικότερα στις κρατικές υπηρεσίες, ο αντίκτυπος ε, των μέτρων που έχουν ε, αναλυθεί για την καταπολέμηση αυτών των φαινόμενων. Υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα αριθμητικά στοιχεία ε, και στατιστικές σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Οι εμπειρογνώμονες θα μας παρουσιάζοντας τις εισηγήσεις τους θα μας δώσουν πολλά τέτοια στατιστικά χρήσιμα στοιχεία. Μετά από αυτή τη σύντομη παρουσίαση θα αφήσω το λόγο στα μέλη του πάνελ, αλλά προ αυτού θα ακούσουμε την συγγήτριά μας, την κυρία Αγγελίλη. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πέρα από τον Πρόεδρο, ευχαριστώ και όλο το προσωπικό του θεματικού τμήματος που διοργάνωσε αυτή τη συνάντηση. Χαιρετίζω τη δόκτωρα Σάμεκ όλους τους παρόντες συναδέλφους και, και τους εισηγητές που θα πάρουν το λόγο. Πρέπει πάντα να ξεκινάμε από τα στατιστικά στοιχεία που αλίμον όσον αφορά την ανεργία και πιο συγκεκριμένα όσον αφορά την ανεργία των νέων ε, είναι ανησυχητικά και συνεχώς αυξάνεται το επίπεδο της ανεργίας. Οι νέοι άνεργοι στην Ευρώπη είναι σχεδόν το 25% ένας νέος τους τέσσερις δεν έχει εργασία στην Ευρώπη και ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι το στοιχείο είναι όσον αφορά εκείνους που είναι νέοι 15 με 24 ετών που εκτός από το ότι είναι άνεργοι είναι και εκτός κάθε κύκλου εκπαίδευσης και κατάρτισης. ΝΕΤ όπως αποκαλούνται. Μιλάμε για 7,5 εκατομμύρια νέους στην Ευρώπη ένας αριθμός ε, πραγματικά εντυπωσιακό αρνητικά. Όπως έλεγε ο Πρόεδρος, πρέπει να ρίξουμε μια ματιά και στη διάσταση του φύλου όταν συζητάμε την ανεργία των νέων. Ας δούμε τα στοιχεία όσον αφορά την απασχόληση των γυναικών, τα σχετικά με τις επισφαλείς ή ευέλικτες μορφές εργασίας, μερικής απασχόλησης ή μη τυπικές μορφές εργασίας και σε αυτούς τους τομείς είναι αρκετά ανησυχητικά τα στοιχεία διότι βλέπουμε ότι η απασχόληση των γυναικών πλήττεται περισσότερο από τα φαινόμενα της επισφαλούς εργασίας και της ευελιξίας. Το τρίτο τρίμηνο του 2012 ανάμεσα στη συνοικία 15-24 με τη μερική απασχόληση, περίπου το 60% από αυτούς ήταν γυναίκες. Δηλαδή η πλειοψηφία των ε, ε, εργασιών, θέσεων εργασίας μερικής απασχόλησης ήταν, ε, εκτελούνται από γυναίκες. Και όσον αφορά τις προσωρινές ορισμένου χρόνου στην τογενή τομέα, πτυχιακές σε πτυχιακό επίπεδο ε, ή μεταπτυχιακό, 64% είναι οι γυναίκες. Ακόμα πιο μεγάλο ποσοστό. Όσον αφορά την κατάρτιση των γυναικών επί της ουσίας, να επενθυμίσω ένα σημαντικό στοιχείο. Το 60% των γυναικών είναι πτυχιούχες. Οι γυναίκες λοιπόν από την έποψη της ε, κατάρτισης ε, σίγουρα θέλουν και πετυχαίνουν ένα ψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθεί να υπάρχει το κενό των φίλων άνηση αμοιβή. Δηλαδή, πολύ συχνά οι γυναίκες κατά μέσο όρο πληρώνονται 17% λιγότερο από τους άντρες για την ίδια εργασία. Αυτούς τους μήνες προσπαθούμε να βρούμε συγκεκριμένες απαντήσεις για, τους, για τις νέες γυναίκες και τους νέους άνδρες, τους ανέργους και τις άνεργες. Δεν θέλουμε να σταματήσουμε αποκλειστικά στα στατιστικά στοιχεία, αλλά θέλουμε να συζητήσουμε και να εντοπίσουμε τις βέλτιστες πρακτικές, τα προγράμματα, τις πολιτικές, τα μέτρα που έδωσαν τα βέλτιστα αποτέλεσματα και θέλουμε να αναλύσουμε αυτά τα στοιχεία, να τα γνωρίσουμε για να τα μοιραστούμε. Να τα διαθέσουμε σε όλα τα κράτη-μέλη αυτά τα στοιχεία, ούτως ώστε τα αποτελέσματα, τα πλέον επιτυχή, να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης. Θέλουμε στην επόμενη προγραμματική περίοδο των κοινοτικών ταμείων, προγραμματισμό 2014 δηλαδή μέχρι 2020, να υπάρχουν αυστηρότερα κριτήρια και ποσοτικοποιημένα κριτήρια όσον αφορά τη χρηματοδότηση, αξιολόγηση και έλεγχο της χρήσης των εθνικών ταμείων και κυρίως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Αυτό γιατί, διότι χρειαζόμαστε την καλύτερη δυνατή χρήση των κοινοτικών πόρων, να χρησιμοποιούνται σε χρήσιμα προγράμματα, να δημιουργούμε ποιοτική κατάρτιση και εκπαίδευση και να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας. Πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιούνται καλύτερα τα κοινοτικά ταμεία. Πιθανότατα θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία, καλύτερος έλεγχος και συντονισμός μεταξύ εθνικών κρατών, κρατών μελών και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μετά θέλουμε να φροντίσουμε ούτως ώστε Πράγματι γίνει αποδεκτό το πρόγραμμα του Youth Employment Initiative και το Youth Guarantee εγγύηση για τους νέους. Και αυτό που θέλουμε είναι να συμμετάσχουν στο μέγιστο βαθμό οι νέοι στην όλη διαδικασία λήψης αποφάσεων για να τους δώσουμε την ορθή αναγνώριση, τη σημασία που πρέπει και να μπορέσουν να πρωταγωνιστήσουν, να τους δώσουμε τη δυνατότητα να συμβάλλουν, να εκφράσουν τις απόψεις τους όσον αφορά τις αποφάσεις που τους αφορούν. Κλείνω λέγοντας ότι οι προτεραιότητες μας είναι η κατάρτιση, η επαγγελματική ποιοτική κατάρτιση. Θέλουμε να ευνοήσουμε την επιχειρηματικότητα, να βοηθήσουμε τους νέους που έχουν μια καλή ιδέα να έχουν πρόσβαση σε πιστώσεις και ενδεχομένως να μελετήσουμε και τρόπους φορολογικής διευκόλυνσης για τους νέους που έχουν καλές ιδέες και που θέλουν να γίνουν επιχειρηματίες, να ακολουθήσουν επιχειρηματική καριέρα. Δεν θέλουμε στους νέους να δώσουμε κάποιες, κάποιους κοινωνικούς μηχανισμούς απόσβεσης. Θέλουμε να δώσουμε ε, μέλλον στους νέους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Αντζελίλη. Θα προχωρήσουμε τώρα στην επόμενη ομιλήτρια, τη Μανουέλα Σάμικ από το IRS. Θα μας παρουσιάσει τις, ε, την κατάσταση των ανέργων νέων ανδρών και γυναικών στην Ευρώπη. Είναι οικονομολόγος που ειδικεύεται στα ζητήματα της αγοράς εργασίας. Από το Μιλάνο, αν δεν κάνω λάθος, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω Ιταλικά μια και είναι η μετρική μου γλώσσα. Ε, Εν πρώτη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε τη δυνατότητα να συμμετάσχω σε αυτό το σεμινάριο και είμαι πολύ ικανοποιημένη που επιτέλους όταν αναλύονται οι τάσεις της αγοράς εργασίας τα πιο πρόσφατα στοιχεία και οι συνέπειες της κρίσεως αρχίζουμε να δίνουμε μεγαλύτερη προσοχή στις διαφορές μεταξύ των φίλων και πιο συγκεκριμένα και όσον αφορά την αγορά εργασίας των νέων, όπως θα δούμε, υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι υπάρχει μια αγορά όπου οι άντρες και οι γυναίκες έχουν τις ίδιες συνθήκες, τις ίδιες δυσκολίες και τις ίδιες ευκαιρίες. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, κυρίως ε, αν θέλουμε να εφαρμόσουμε αποτελεσματικές πολιτικές. Υπάρχει αυτή η προσοχή στα πλαίσια της Επιτροπής Γυναικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχει και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έκανε μεγάλη μελέτη όσον αφορά αυτά τα θέματα και είναι καθοδόν προς ολοκλήρωση η μελέτη. Επιτέλους ξαναμπαίνουμε να μπαίνουμε στην ουσία της διαφοράς των φύλων και χάρη στο γεγονός ότι επιτέλους υπάρχουν στοιχεία, στατιστικά στοιχεία που μας επιτρέπουν να προβούμε σε ενδελεχέστερες αναλύσεις, λεπτομερέστερες αναλύσεις. Στόχος μου σήμερα είναι να κάνω μια παρουσίαση εν συντομία κάποιων ε, βασικών διαφορών που αντιμετωπίζονται και διαπιστώνονται όταν αναλύουμε ποια είναι η συνθήκη για τους νέους στην αγορά εργασίας, κυρίως τις συνέπειες που έχει η κρίση. Λοιπόν, ε, ε, το πρώτο στοιχείο δεν θα μπορέσω να περιγράψω τα πάντα. Το πρώτο, το πρώτο που θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι το εξής, ότι αυτή η κρίση ε, έπληξε περισσότερο τους νέους άντρες από ότι τις νέες γυναίκες. Η απασχόληση των ε, νέων γυναικών μειώθηκε πιο δραστικά, πιο δραστικά ε, ε, αυξήθηκε πολύ πολύ ανεργία των ε, νέων γυναικών. Αν βλέπετε τα στοιχεία όσον αφορά τα επίπεδα της ανεργίας στην πρώτη, στο πρώτο γράφημα που βλέπετε στα αριστερά, βλέπετε το ποσοστό της ανεργίας των νέων 15 μέχρι 24 των ανδρών που είναι πιο υψηλό ποσοστό από αυτό των γυναικών. Όμως όταν αναλύουμε αυτές τις τάσεις θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή διότι ένας δείκτης κατά την άποψή μου πιο πλήρης, πιο εξαντλητικός όσον αφορά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι στην αγορά εργασία δεν είναι τόσο το ποσοστό της ανεργίας αλλά πάνω απ' όλα το net rate, το καθαρό ποσοστό που ανέφερε η κυρία Αντζελίλη. Δηλαδή που λαμβάνει όχι μόνο υπόψη τους νέους που ψάχνουν να βρουν δουλειά, αλλά και τους νέους που δεν ψάχνουν να βρουν δουλειά, που είναι αδρανείς, αλλά δεν είναι ούτε φοιτητέ, ούτε τελούν υποκατάρτιση. Είναι οι νέοι οι οποίοι έχουν βγει εντελώς εκτός της αγοράς εργασίας, που δεν δοκιμάζουν καν να μπουν στην αγορά εργασίας. Είναι οι πιο απόμακροι από την αγορά εργασίας. Άρα αυτοί που κινδυνεύουν περισσότερο με αποκλεισμό από τη δουλειά κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Εάν δούμε αυτό το σύνολο, όπως βλέπετε, από τα δύο άλλα γραφήματα, τα τελευταία, το ποσοστό, η διαφορά μεταξύ το, το καθαρό για τις γυναίκες και μεταξύ νέων και μεγαλύτερων είναι πιο υψηλό της ανεργίας από αυτό των ανδρών. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα κορίτσια πολύ πιο εύκολα είναι αδρανή μετά από κάποιο χρόνο δεν ψάχνουν να βρουν ε, δουλειά και βγαίνουν εντελώ από την αγορά εργασία. Ένα δεύτερο σημαντικό στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι το εξή. Ζητώ συγγνώμη. Α, υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ χωρών και μας δείχνει αυτό ότι εν μέρει αυτές οι διαφορές μπορούν να οφείλονται και στο ε, διαφορετικό αντίκτυπο που έχει η κρίση στις διάφορες χώρες, όμως μπορεί να οφείλονται στο διαφορετικό είδος πολιτικών που εφάρμοσαν οι διάφορες χώρες για να υποστηρίξουν την απασχόληση των νέων. Όπως βλέπετε, οι χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά των νέων, δηλαδή των νέων που είναι εντελώς εκτός παιδείας, κατάρτισης, αγοράς εργασίας, είναι οι σκανδιναβικές χώρες και οι χώρες κεντρικής Ευρώπης. Ενώ οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, της ε, ε, Νότιας Ευρώπης και των Αγγλοσαξονικών χωρών έχουν επίπεδα ποσοστά νέων εκτός των πάντων μεγαλύτερο. Είναι πρόβλημα παρέμβασης και προσοχής που δίδεται στις διάφορες πολιτικές για υποστήριξη της ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας. Υπάρχουν και μεγάλες διαφορές μεταξύ χωρών, όπως θα δούμε υπάρχουν διαφορές φύλου σε αυτό το ποσοστό των net rates. Αυτό που είναι εντελώς εκτός. Σε κάποιες ε, χώρες το ποσοστό ε, net είναι πιο ψηλό μεταξύ των νέων ανδρών, ενώ σε άλλες χώρες είναι πολύ πιο υψηλό ε, στις νέες γυναίκες. Το net, αυτό που είναι εντελώς έξω από αγορά εργασίας, παιδεία, κατάσταση κλπ. Άλλη σημαντική διαφορά ε, που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι κάτι που το ανέφερε ήδη, αναφέρθηκε ήδη. Η διαφορετική σύνθεση αυτού του πληθυσμού. Ενώ ανάμεσα στα, στους άντρες οι περισσότεροι νετ είναι οι νέοι οι άνεργοι, οι νέοι που ψάχνουν να βρουν δουλειά, ενώ στις ε, γυναίκες οι περισσότεροι ε, περισσότερες είναι οι αδρανεί γυναίκες, τα αδρανή κορίτσια που δεν ψάχνουν κάμια δουλειά. Αυτή η συνιστόσα, η αδρανής, ούτε παιδεία, ούτε, ούτε εκπαίδευση, ούτε κατάρτιση αυξάνεται με την αύξηση τη ηλικία. Είναι πολύ πιο υψηλό το ποσοστό στα κορίτσια ανάστα 25 με 29 από ότι για τα κορίτσια από 14 μέχρι 24 γιατί πιθανότατα είναι ένα φαινόμενο που συνδέεται με το γεγονός ότι από τα 25 μέχρι 29 τα κορίτσια αρχίζουν να έχουν οικογένεια, να έχουν παιδιά και είναι πολύ πιο δύσκολο για αυτές να παραμείνουν στην αγορά εργασίας. Ήδη λοιπόν εδώ διαφαίνεται ένα στοιχείο, δηλαδή ότι τα προβλήματα που συνδέονται με την συμφιλίωση εργασιακής ζωής και οικογενειακής ζωής αρχίζει να διαφαίνεται ήδη σε νεανική ηλικία και αυτό ίσως να αφήνει διαχρονικά αποτελέσματα. Αν νέοι είναι εκτός της αγοράς εργασίας θα είναι πολύ πιο δύσκολο να ε, ξανά ενταχθούν όσο ενταχθούν στην αγορά εργασίας όσο αυξάνεται η ηλικία. Άρα έχουμε διαφορετικό αντίκτυπο της αδράνειας όσον αφορά την απασχόληση μεταξύ νέων γυναικών και νέων ανδρών. Και αυτό το βλέπουμε και αν κοιτάξουμε ποιες διαφορές υπάρχουν όσον αφορά τους λόγους για τους οποίους οι γυναίκες δηλώνουν ότι είναι αδρανείς, ανενεργές, εν συγκρίση με τους άντρες. Ενώ ανάμεσα στις νέες κοπέλες ο λόγος, ο βασικός είναι οικογενειακή, το οικογενειακό φορτίο, περίπου 50% των νέων γυναικών, ναι, των αδρανών λένε ότι είναι έτσι λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων, ενώ στους νέους άντρες ούτε το 7% δεν το λέει αυτό. Η αποθάρρυνση όμως είναι πολύ πιο μεγάλη ανάμεσα στους νέους άντρες σε σύγκριση με τις νέες γυναίκες. Η αδράνεια για τις κοπέλες οφείλεται περισσότερο σε οικογενειακές υποχρεώσεις, όσον αφορά τους νέους άντρες οφείλεται περισσότερο στην αποθάρρυνση, απογοήτευση. Δεν μπαίνω στην ουσία των διαφορών λόγω εκπαίδευσης για άλλα χαρακτηριστικά προσωπικά διότι στις επόμενες παρεμβάσεις ε, πιθανότατα θα υπάρξει βάθυνση σε αυτές τις πτυχές. Θα ήθελα να αναφερθώ στο ότι είναι σημαντική εκπαίδευση, το επίπεδο για τις νέες κοπέλες. Τα... Η συνέπεια ε, ε για αυτές που έχουν επιτυχία πανεπιστημιακά ε, είναι πολύ πιο χαμηλά τα ποσοστά εκείνων που είναι εντελώ εκτό. Αλλά υπάρχουν συγκεκριτικά στοιχεία σε κάποιε χώρε τη ε, Μεσογειακή Ευρώπη, όπω είναι η Ιταλία, όπου εκεί αυξάνεται και κατά πολύ η έξοδο από την αγορά εργασία από κοπέλε που έχουν πτυχία υψηλού επίπεδου. Εδώ υπήρχε το γράφημα, όμως νομίζω ότι δεν βλέπουμε πολύ καλά δυστυχώς, όπου εκεί κανονικά θα βλέπατε τα ποσοστά στο πιο διαφανές ανοιχτό κομμάτι του διγραφήματος ανδρών και γυναικών που είναι ανενεργοί σε σχέση με τους ε, ανέργους. Περισσότερο ανεργία από ότι ανεργοί. Όσον αφορά τις οικογενειακές υποχρεώσεις, σαν εξήγηση της εξόδου αγορά εργασία, βλέπετε εδώ στο γράφημα, ε, γίνεται σύγκριση, σύγκριση των ποσοστών των νέων, των ανδρανών, των ανενεργών ε, που δεν είναι στην κατάρτιση εκπαίδευση, σύγκριση μεταξύ ανδρών και γυναικών. Κάνουμε σύγκριση μεταξύ εκείνων που έχουν παιδιά και εκείνων που δεν έχουν παιδιά. Και βλέπετε ανάμεσα στι κοπέλε, αυτέ που έχουν παιδιά είναι οι πιο ανοιχτέ ε, γραμμέ του ιστογραφήματο. Ανάμεσα στι κοπέλε που έχουν παιδιά, το ποσοστό των net, των αδρανών, είναι πολύ πιο υψηλό σε σχέση με τι κοπέλε που δεν έχουν παιδιά. Ε, για μία ακόμη φορά, βλέπουμε τι οικογενειακέ υποχρεώσει που είναι μια σημαντική εξήγηση. Λοιπόν, Λοιπόν, για να σας αγαπώ κάποια συμπεράσματα. Ποιες είναι οι βασικές συνιστώσεις των διαφορών όσον αφορά τη συμπεριφορά και τη στάση όσον αφορά την αγορά εργασίας και ανάμεσα στους νέους. Όταν κανείς θα περίμενε μικρότερες συνέπειες. Πρώτο πρόβλημα που είδαμε καθαρά αφορά τα θέματα φροντίδας και το άλλο αφορά και το διαχωρισμό που υπάρχει όσον αφορά την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ένα από τα προβλήματα που διαφαίνεται από τα στοιχεία αλλά και τις μελέτες που διενεργήθηκαν όσον αφορά αυτά τα ζητήματα είναι το εξή. Οι κοπέλες τείνουν να έχουν είδος κατάρτισης που είναι πιο δύσκολο μετά να, βρει, να βρουν δουλειά στην αγορά εργασίας. Οι κοπέλες τείνουν να έχουν επίπεδα εκπαίδευσης που δεν ανταποκρίνονται, δεν, ε, ε, δίνουν τι δεξιότητε που απαιτούν οι επιχειρήσει και αγορά εργασία, άρα δυσκολεύονται περισσότερο οι κοπέλε αυτέ να βρουν δουλειά. Και οι κοπέλε επιπλέον ε, εμπλέκονται λιγότερο στην κατάρτιση, κυρίω και στι πληροφορίε όσον αφορά τη εργασία Στο ΣΕΝΤΕΦΟ που έκανε μια μελέτη όπου διαφαίνονται αυτέ οι διαφορέ πάρα πολύ ξεκάθαρα. Ε, τρίτο πρόβλημα είναι τα στερεότυπα και οι διακρίσεις που υπάρχουν όσον αφορά τις αποφάσεις για την πρόσληψη σε επιχειρήσεις και τις αποφάσεις για μείωση προσωπικού. Και εδώ υπάρχει αυτό το στοιχείο που κατά την άποψή μου είναι εμβληματική σημασία που διαφαίνεται και απόρρεα από το τελευταίο ευρωβαρόμετρο που παρουσιάστηκε εδώ ε, πριν από καιρό όπου διαφαίνεται σαφώς ποια είναι η αντίληψη, τα κριτήρια που υιοθετούν οι επιχειρήσεις όταν αποφασίζουν προσλήψεις και όπως ε, θα βλέπετε υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ των κριτηρίων που, θεω, που ισχύουν για την πρόσληψη των γυναικών σε σύγκριση με τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την πρόσληψη ανδρών. Για τους άντρες η επαγγελματική εμπειρία, το επίπεδο των γνώσεων, η ευελιξία, όσον αφορά το ωράριο εργασία είναι πολύ πιο σημαντικά από ό,τι για τι γυναίκε. Ενώ οι γυναίκε σε πρώτη θέση είναι το αν έχουν ή δεν έχουν παιδιά. Για μία ακόμη φορά τα θέματα φροντίδα παραμένει ευελιξία όσον αφορά το ωράριο εργασία. Αλλά υπησέρχεται και η φυσική πτυχή, η φυσική ουσιαστικά. Όσον αφορά τα προσόντα επαγγελματική εμπειρία, αυτά έχουν πολύ μεγάλη, λιγότερη σημασία για τις γυναίκες. Τέταρτο σημαντικό στοιχείο που μπορεί να εξηγεί τις διαφορές μεταξύ νέων στην αγορά εργασίας είναι και τα αποτελέσματα της πολιτικής εργασίας, των διαφόρων συστημάτων ρύθμισης αγοράς εργασίας, των πολιτικών υποστήριξης για, τις, για την εργασία περίθαλψης και υποστήριξης και φροντίδας που μέχρι τώρα χαρακτηρίζονται από πολύ χαμηλό επίπεδο προσοχής είναι λιγότερο αποτελεσματικά τα μέτρα αυτά όσον αφορά τι γυναίκε. Δεν λαμβάνουν υπόψη επαρκώ τι αφορά το φύλλο. Στη μελέτη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχει μια ανάλυση όσον αφορά τι διάφορε παρεμβάσει με το φύλλο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο. Παρεμβάσει που έγιναν τα τελευταία χρόνια για την υποστήριξη απασχόληση των νέων. Και πολύ συχνά ε, λείπει η προσοχή στι διαφορέ των φύλων. Και κλείνω. Ποιες είναι οι συνέπειες της ανεργίας των νέων αλλά και της πολύ μικρής προσοχής που δίδεται στις διαφορές των φύλων. Και εδώ ε, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη τεκμηρίωση και στοιχεία επιστημονικά που δείχνουν ότι το πέρασμα το σχολείο στη δουλειά είναι μια περίοδος πάρα πολύ ευαίσθητη και αυτό που συμβαίνει κατά τη διάρκεια αυτής της μετάβασης κινδυνεύει να επηρεάσει τους όρους ζωής, ε, το εισόδημα και την υγεία των ατόμων καθ' τα επόμενα χρόνια. Μιλάμε για το scaring effect, scarring effect, δηλαδή ότι αφήνει κάποια ουλή το πρόβλημα αυτό. Όταν υπάρχει πρόβλημα ανεργία στην αρχή της εργασιακής ζωής, ίσως να έχει μόνιμο αντίκτυπο, μακροχρόνιο. Αφήνει ουλέ και μπορεί να αρνητικέ συνέπειε για τι γυναίκε, διότι νέε γυναίκε, όπω είδαμε, βγαίνουν ε, εντελώ από την αγορά εργασία επί μακρά περίοδο. Ποιε είναι αυτέ οι συνέπειε μεγάλη κίνδυνη, μεγαλύτερη κίνδυνη φτώχειας και μείωσης των προοπτικών απασχόλησης, εισοδήματος κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Αυτό και πάνω απ' όλα διότι τα τελευταία χρόνια και η μεταρρύθμιση των συστημάτων του κράτους προνοίας, η μεταρρύθμιση των εξαιρετικών συστημάτων συνδέουν πιο στενά όλο και πιο στενά το μελλοντικό εισόδημα, τα συνδιοξιδετικά ευεργετήματα με τι συνεισφορέ που καταβάλλονται κατά τη διάρκεια τη εργασιακή ζωή. Εάν είναι κατακαιρματισμένη η εργασιακή ζωή, δεν είναι συνεχή με μακρά περιόδου εκτό αγορά εργασία, αυτό σημαίνει ότι μετά, σαν ηλικιωμένοι, αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν πιο χαμηλή σύνταξη. Άρα αυξάνεται ο κίνδυνο φτώχεια. μικρότερη πρόσβαση στην κοινωνική προστασία. Σε πολλέ χώρε μπορεί κανεί να έχει επίδομα ανεργίας και διάφορες μορφές κοινωνικής προστασίας, όμως αν υπάρχει ένα είδους εργαστικής εμπειρίας, αν δούλεψε κανείς τουλάχιστον μια χρονική περίοδο, αν εργάζεται επί συγκεκριμένο αριθμό ωρών κλπ. Το είναι κανείς εκτός αγοράς εργασίας σημαίνει να έχει και μικρότερες δυνατότητες πρόσβασης στην κοινωνική πρόνοια. Τρίτο πρόβλημα είναι ότι σπαταλώνται πόροι. Αναφέρθηκε και πριν μάλλον πόροι, ε, ταλέντα. Οι γυναίκες έχουν περισσότερα προσόντα από τους νέους και το, όταν οι κοπέλες εκτός αγοράς εργασίας η κοινωνία ε, σπαταλά ταλέντος, σπαταλά πόρους. Το κόστος δεν είναι μόνο κόστος ατομικό, αλλά είναι και κόστος κοινωνικό. Ε, δύο στοιχεία θα ήθελα να σας δείξω. Α, τελείωσα, ναι, ναι. Βλέπουμε δίκτυο κινδύνου φτώχειας ποσοστό νέων από 18 μέχρι 24 ετών που κινδυνεύουν να πέσουν στη φτώχεια ή να πέσουν σε κοινωνικό αποκλεισμό. Η τάση από το 2005 μέχρι το 2011 βλέπετε Ποιο είναι. Η κόκκινη γραμμή είναι οι κοπέλες έχουν κίνδυνο φτώχειας πιο υψηλό από ότι οι νέοι. Οι νέοι έχουν κίνδυνο και εν γέννη οι νέοι έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχεια από ότι οι ενήλικε, οι μεγαλύτεροι. Όσον αφορά την πρόσβαση στην κοινωνική πρόνοια. Έχουμε εδώ στοιχεία που καταδεικνύουν ότι οι νέες σε σχεδόν όλες τις χώρες το ποσοστό των νέων γυναικών που λαμβάνει ενίσχυση είναι πολύ πιο χαμηλό από τους νέους ακριβώς διότι οι νέες είναι εκτός της αγοράς εργασίας άρα δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μια ολόκληρη σειρά μηχανισμών κοινωνικής προστασίας και πρόνοιας που όμως είναι διαθέσιμη για εκείνους που είναι μέσα στην αγορά εργασίας. Λοιπόν, για να κλείσω, οι διαφορές του φίλου, των φίλων, ήδη διαπιστώνται σε νέα ηλικία όταν μπαίνει κανείς στην αγορά εργασίας. Το γεγονός ότι οι νέες έχουν μεγαλύτερες δυσκολίες και μεγαλύτερη πιθανότητα να βγουν εξ ολοκλήρου από την αγορά, καθιστά τον κίνδυνο φτώχειας τον κίνδυνο αποκλεισμού κατά τη διάρκεια της ζωής τους πολύ πιο υψηλό. Και αυτό σημαίνει ότι οι διαφορές των φύλων πρέπει να αντιμετωπίζονται από την αρχή στα πλαίσια των πολιτικών με πολιτικές που τείνουν να λαμβάνουν υπόψη αυτές τις διαφορές. Οι δεμοί δεν είναι αποτελεσματικές. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σαμίκ. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την εξαιρετική εισαγωγή και τις ε, σχετικές πληροφορίες για το θέμα μας και πιστεύω πως πραγματικά τονίσατε σαφέστατα ότι υπάρχουν διαφορές ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες σε πολλούς τομείς. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πολύ γι' αυτό. Θα συνεχίσουμε τώρα με ορισμένες ερωτήσεις, αλλά πρώτα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Γυναικών, την κυρία Μόριν Σαχτιέ θα λάβει το λόγο γιατί είναι η συγγήτρια μιας έκθεσης ε, με τίτλο η επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην ισότητα και τα δικαιώματα των γυναικών» και θα μας δώσει μερικές ε, πληροφορίες από το Ευρωβαρόμετρο. Ε, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Merci, Merci. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τη Ρομπέρτα, την Αντιπρόεδρό μας για τη διοργάνωση της σημερινή ακρόασης για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα για το οποίο πιστεύω ότι και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο δεν υπάρχει μια επαρκή κινητοποίηση σε σχέση με το, την, το μέγεθος του προβλήματος και τη διαχρονικότητά του, διότι το είπατε κι εσείς, ότι ό,τι σπέρνουμε σήμερα θα το οργώσουμε για πολλές γενιές ε, στη συνέχεια. Ε, στον απόϊχο της δικής σας παρέμβασης και ας μην ξεχνούμε ότι χρησιμοποιήσαμε συγκρίσιμες πηγές δεδομένων, θα έλεγα τα εξής. Πρώτα απ' όλα, ε, ήδη στο σχολείο ε, υπάρχει μια ουσιαστική διακριτική μεταχείριση. Εσείς μιλήσατε για προσανατολισμό, δεν επανέρχομαι, συμφωνώ μαζί σα. Πέραν αυτού, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι υπάρχει και ένα άλλο είδο διακριτική μεταχείρισης. Όταν μιλάμε για έλλειψη δεξιοτήτων ε, στα συστήματα κατάρτιση, είναι σε δυσμενέστερη θέση τα κορίτσια. Γιατί, διότι σε σχέση ε, με τα αγόρια και αν δεν ακολουθήσουν ε, μια πιο ε, προχωρημένη εκπαίδευση, εγκαταλείπουν νωρίτερα από τα αγόρια. Ελπίζω να με παρακολουθείτε. Ε, και όταν μιλήσατε για τα συστήματα κατάρτισης ότι όταν υπάρχουν ναι, προβλήματα, δημιουργούν και περισσότερα προβλήματα τα αγόρια και εγκαταλείπουν ε, νωρίτερα από τα κορίτσια. Ενώ τα κορίτσια ε, παραμένουν ε, μέσα στο σύστημα, δεν αντιδρούν τόσο βία, όμως δεν έχουν μια καλή έκβαση και αυτό ε, εν τέλει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπατε σε σχέση με τον προσανατολισμό που επιλέγουν τα δύο que... Κάτι άλλο εξίσου σημαντικό ε, είπαμε ότι η κατάρτιση αγοριών και κοριτσιών ε, είναι περίπου εισάξια σήμερα. 70% των κοριτσιών έχουν ε, πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Είτε μιλάμε για την ιατρική, για την υγεία γενικότερα στο δίκαιο, στην νομική. Έχουν αντίστοιχες επιδόσεις, αλλά υπάρχει διαφορετική μεταχείριση. Δεν είναι φιέστερα τα κορίτσια. Δεν εννοώ αυτό, αν και υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι μαθαίνουν την ανάγνωση ένα χρόνο νωρίτερα από τα αγόρια. Ε, δέχονται καλύτερα το, τη λειτουργία του συστήματος ε, κατάρτισης. Λοιπόν, τα συστήματα κατάρτιση λειτουργούν και με ιδιωτικέ, αλλά και με κρατικές επενδύσεις. Επενδύσεις από πλευρά του κράτους και από πλευρά των νοικοκυριών. Τι, τι περιμένουμε, πώς χρησιμοποιούμε αυτές τις επενδύσεις που κάνουμε. Η κρίση μας κατέδειξε ότι καθυστερεί περισσότερο ο είσοδο των κολλησιών στην αγορά εργασία. Έξι μήνες περισσότερο κατά μεσόωρο χρειάζονται για να ε, καταλάβουν την πρώτη θέση απασχόλησης. Κατά την πρόσληψη υπάρχει διακριτική μεταχείριση, αυτό το αποδείξατε με τα στοιχεία σας και βάσει αυτό που μας είπατε συνεχίζω και εγώ ένα λεπτάκι να δούμε, βλέπουμε και τις διαφάνειες ταυτόχρονα. Ας δούμε τα κριτήρια για την πρόσληψη. Θέλω να το δείτε διότι μου φαίνεται απίστευτο τη σήμερον ημέρα. Συχνά σχολιάζω αυτό το ζήτημα στις ε, διασκέψεις για το ζήτημα αυτό και δεν με πιστεύουν όταν τα λέω. Το πρώτο κριτήριο για μια γυναίκα είναι έχετε παιδιά, ή είστε στην ε, ε, κατάλληλη ηλικία ή, έχετε, ή σκοπεύετε να αποκτήσετε παιδιά. Αυτό είναι το πρώτο κριτήριο. Ε, κατά πόσο είστε διαθέσιμοι ως προς τα ευέλικτα ωράρια εργασίας. Αυτό είναι το δεύτερο κριτήριο. Για την επαγγελματική εμπειρία δείτε στην αριστερή στήλη ε, είμαστε στην 7η θέση ως προς τα κριτήρια πρόσληψης. Ενώ σας είπα ότι το 70% των πτυχιούχων ε, ε, είναι από το γυναικείο φύλλο. Άρα οι επενδύσεις που έγιναν, ιδιωτικές και κρατικές, οδήγησαν σε αυτό το 70%. Στην πρόσληψη όμως αυτό το κριτήριο είναι στην 7η θέση. Τι συμβαίνει τώρα για, στην περίπτωση των αντρών. σκεφτείτε ότι αυτό αφορά τα παιδιά σας ή τα εγγόνια σας ε, και δεν θα χαμογελάτε τόσο πολύ όταν θα σας εξηγήσω τι συμβαίνει. Ε, βλέπουμε τα κριτήρια λοιπόν για τους άντρες. Στη δέκατη θέση είναι η ερώτηση για τα παιδιά και όχι στην πρώτη. Οι γυναίκες λοιπόν με δεξιότητες που έχουν πανεπιστημιακά πτυχία κατά την πρόσληψη δεν μπορεί να χρησιμοποιήσουν αυτό το ατού που έχουν. Αυτά βασίζονται σε βιώματα, σε μαρτυρίες. Οι γυναίκες το γνωρίζουν πολύ καλά ότι κατά την πρόσληψη η εξωτερική εμφάνιση έχει ιδιαίτερη σημασία. Είναι στην τρίτη θέση αυτό το κριτήριο. Δείτε αυτή την ε, ε, γραφική παράσταση. Βλέπουμε το μέσο όρο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αριστερά, ως προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, βλέπετε χώρες όπου είναι ιδιαίτερα αισθητή η διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλλα για τα κριτήρια της πρόσληψης πάλι συγκεκριμένα το πρώτο για τις γυναίκες, ε, δηλαδή αν έχουν παιδιά ή όχι, συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, ε, αυτός είναι ένας τομέας όπου πρέπει να δράσουμε κατά προτεραιότητα, διότι είναι ένας από τους μεγαλύτερους φραγμούς ε, κατά την πρόσληψη. Δεξιά τώρα, όσο προχωρούμε προς τα δεξιά, βλέπουμε μειούμενη την διαφορά όπως βιώνεται, τονίζω αυτό, από τους ενδιαφερόμενους και τις ενδιαφερόμενες. Ε, αν δούμε τις διαφορές ε, στην Κύπρο και τη Βουλγαρία, παραδείγματος χάρη, εκεί δεν ε, χρησιμοποιείται αυτό το κριτήριο κατά την πρόσληψη επίσημα, αλλά το ζουν έτσι οι γυναίκες. Το ευρωβαρόμετρο χαρτογραφεί αυτή την κατάσταση με συγκεκριμένα στοιχεία και άρα έχουν σημασία τα αριθμητικά στοιχεία που λαμβάνουμε από το ευρωβαρόμετρο. Τρίτη γραφική παράσταση, εδώ βλέπετε τις διαφορές στην πρόσληψη των δύο φύλων. Διαπιστώνεται ότι είναι αντίστροφες οι τάσεις. Σε ποιο κριτήριο προσδίδει ο εργοδότης μεγαλύτερη σημασία ανάλογα με το φύλλο. Εκεί βλέπετε πως η επαγγελματική εμπειρία έχει πολύ μεγαλύτερο ειδικό βάρος για τους άντρες σε σχέση με τις γυναίκες. Λοιπόν, τα νέα κορίτσια ε, ολοκληρώνουν σπουδές τους αργότερα χωρίς τόσες πολλές δεξιότητες. Ε, καθυστερούν περισσότερο για να βρουν την πρώτη θέση απασχόληση παρότι έχουν περισσότερα πτυχία ή περισσότερες επαγγελματικές δεξιότητες γιατί έχουν, είναι σε δυσμενέστερη θέση ως προς τα κριτήρια πρόσληψης. Α, και παρέλειψα κάτι πολύ σημαντικό. Το θέμα της διαθεσιμότητάς τους για το ωράρια εργασίας λόγω των παιδιών ακριβώς. Να άλλο ένα κριτήριο αρνητικής διακριτικής ε, μεταχείρισης Πέραν αυτού υπάρχει η χαμηλότερη αμοιβή. Τα νεαρά κορίτσια προσλαμβάνονται με χαμηλότερο μισθό κατά μέσο όρο κατά 16,7% και για να προσθέσουμε και το κερασάκι σαν να μας έφταναν όλα αυτά με κάθε ε, νέα γένα βάσει στοιχείων του ΩΣΑ με κάθε γένα έχουμε μία μισθολογική διαφορά ανάμεσα στα δύο που ανέρχεται στο μείον 12% κατά των γυναικών, δηλαδή χαμηλότερος μισθός κατά 12%. Άρα δεν είναι τόσο μεγάλο το ε, μισθολογικό θέλγητρο. Πέρα από τα προβλήματα της συμφιλίωσης της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής, σε συνδυασμό και με την οικονομική κρίση, οι γυναίκες που απασχολούνται μερικώς, διότι αυτή είναι μια διέξοδος ε, για τις γυναίκες ε, ε, για να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα προβλήματα που προανέφερα. Απασχολούνται λοιπόν μερικώς, όπως είπα, εκείνες ε, σιωπηρά απέρχονται από αυτήν την αγορά εργασίας ε, διότι δεν βρίσκουν άλλη διέξοδο και υφίστανται άμεσα τον αντίκτυπο της κρίσης και ε, ε, εξ πρωτοβουλίας ε, εξέρχονται από την επίσημη αγορά εργασίας και ασχολούνται με θελοντικές δραστηριότητες οδηγούμενες έτσι στην Θα σταματήσω εδώ γιατί πρέπει να είμαι και σύντομη. Δεν νομίζω να έχουμε και περισσότερο χρόνο, Πρόεδρε, αλλά ήθελα κλείνοντας να σας πω ότι θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση σε σχέση με αυτό το πρόβλημα όλος ιδιαίτερο της φτωχοποίησης των γυναικών είναι οικονομικού, πολιτικού και κοινωνικού χαρακτήρα αυτό το πρόβλημα. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Μογάν Σαχτιέ. Όπως σας είπα και στην αρχή, η κυρία Μογάν Σαχτιέ είναι ήταν η συγγήτρια για μια πολύ σημαντική ε, έκθεση για την οικονομική κρίση που ενεκριθεί στην Ολομέλεια το Μάρτιο ε, και πραγματευόταν τις επιπτώσεις κρίσης ε, ε, στα δύο φίλε. Εργαστήκατε πάρα πολύ σκληρά για αυτό το ζήτημα και σας ευχαριστούμε που ήρθατε ε, στη σημερινή μας ακρόαση. Θα ήθελα τώρα να αρχίσει το στάδιο των ερωταπαντήσεων, ε, να ακούσουμε τους βουλευτές και όχι μόνο, αν έχουν να ρωτήσουν κάτι. please. Thank you very much for organizing this and the uh, two presentations. They were... Ευχαριστώ πολύ καταρχάς για τη διοργάνωση. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το σημερινό σεμινάριο. Θα ήθελα να ρωτήσω σε γενικέ γραμμέ τι έχετε βρει όσον αφορά τι περιφερειακέ διαφορέ. Εγώ είμαι από την Ουγγαρία, μια χώρα, νέα χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με κομμουνιστικό παρελθόν και πάντα με σοκάρει και με ενοχλεί το γεγονό ότι κάνουμε λόγο για ζητήματα απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά. Είναι λίγο καλύτερο να μιλήσουμε τουλάχιστον για τα ζητήματα της, ε, ε, του φύλου, αλλά θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για, γεωγραφι... για τις γεωγραφικές πτυχές, για τις πολιτικές πτυχές, ε, Ανατολική Ευρώπη σε σχέση με τη Δυτική Ευρώπη. Ποιες είναι οι διαφορές που έχετε βρει εκεί και τι θεωρείτε θετικό από την άποψη της γυναικείας κινητικότητας. Άλλο βέβαια είναι η θεωρία, αλλά στην πράξη η κινητικότητα των γυναικών είναι κάτι το δυσάρεστο, είναι εξαναγκαστική μετανάστευση. Οι γυναίκες αυτές αναγκάζονται να αφήσουν τον τόπο τους, τη χώρα τους, την πατρίδα τους και τις οικογένειές τους πολλές φορές πίσω και να μεταναστεύσουν σε χώρες όπου πολλές φορές αναγκάζονται να κάνουν ε, πολύ κακοπληρωμένες δουλειές, ε, οικιακές βοηθοί για παράδειγμα, καθαρίστριες ε, σε πλουσιότερες χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Έχουν διεξανθεί μελέτες για αυτό το θέμα ή έχετε κάποιο έβριγμα σχετικά με αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία. Κυρία Σάμεκ, θα θέλατε να απαντήσετε. Ναι, υπάρχουν διαφορές μεταξύ χωρών αρκετά σημαντικές όσον αφορά όλους τους ε, δείκτες και αυτό που φαίνεται να γίνει στις χώρες Ανατολικής Ευρώπης ε, και σε κάποιες κυρίως οι διαφορές μεταξύ των φύλων και η επιδείνωση της θέσης των γυναικών ε, είναι ιδιαίτερα μεγάλα, μεγάλη και το φαινόμενο της μετανάστευσης. Οι γυναίκες σαν ε, πρώτοι μετανάστες που μετά υποστηρίζουν την οικογένεια στη χώρα τους με τη δουλειά που κάνουν σε άλλες χώρες. Και αυτό είναι ένα φαινόμενο πολύ ε, σημαντικό. Υπάρχουν μελέτες. Μελέτες που έγιναν στην Ιταλία κυρίως όσον αφορά ε, εκείνων που είναι περιπλανόμενοι όπως λέμε. δηλαδή που προσφέρουν τη δουλειά περίθαλψης υπηρεσίες περίθαλψης κυρίως για τους ηλικιωμένους. Δεν είμαι σε θέση να σας παρουσιάσω συγκεκριμένα στοιχεία, αλλά λυθεύει. Υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές σε εθνικό επίπεδο. Υπάρχουν διαφορές και στα μεταναστευτικά φαινόμενα, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση κρατή για τις γυναίκες μετανάστριες. Και αυτό αυτό είναι ενδιαφέρον διότι αλλάζει και το είδος και ο τρόπος μετανάστευσης. Πριν μετανάστευαν οι άντρες, τώρα μεταναστεύουν περισσότερο οι γυναίκες και αυτό επηρεάζει τις οικογένειες, τα παιδιά που εγκαταλείπονται στη χώρα καταγωγής ε, και τελικά κινδυνεύουν να φτωχύνουν οι χώρες ε, προέλευσης. Δεν έχω όμως ε, κάποια συγκεκριμένα στοιχεία να σας δώσω για να τα υποστηρίξω αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κλεβέτη. Θα μιλήσω ρουμανικά. Θα ήθελα να κάνω ορισμένα σχόλια. Θα είμαι σύντομη γιατί πρέπει να πάω σε ψηφοφορία στην Επιτροπή Απασχόλησης. Λοιπόν, για μένα το πιο σημαντικό ζήτημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να βρούμε λύση είναι τα στερεότυπα. Άκουσα την παρουσίαση της κυρίας Μωράν Σαχτιέ και μπορώ να σας πω ότι πραγματικά με λυπεί που άκουσα αυτά τα πράγματα. Είναι αλήθεια και αληθεύουν για ποιους λόγους. Καταρχάς υπάρχει κοινωνική πίεση προς τις γυναίκες για να κάνουν παιδιά. Οι γεννήσεις μειώνονται και τα παιδιά λιγοστεύουν. Όμως οι γυναίκες ταυτόχρονα πρέπει να εργαστούν κιόλα. Έχουν σπουδάσει και ζούμε στον 20ο αιώνα. Εάν δεν δουλεύουμε δημιουργούνται ερωτηματικά. Πώς δηλαδή κερδίζουμε τα προστοζήν. Επίσης υπάρχει η πίεση της συμφιλίωσης εργασίας και οικογένειας. Βέβαια η οικογένεια απαιτεί αφιέρωση πολλού χρόνου έπειτα υπάρχουν και τα στερεότυπα, τα στερεότυπα των ρόλων. Τι ρόλο έχει αναλάβει μια γυναίκα, τι ρόλο έχει αναλάβει ένα άντρα. Είναι πολύ δύσκολη η συμφιλίωση οικογένειας και καριέρας και αυτός ο ρόλος πέφτει συνήθως στα χέρια των γυναικών. Πολλές φορές ε, πραγματικά έχω την εντύπωση ότι οι γυναίκες είναι παγιδευμένες σε έναν ιστό αράχνης, πρέπει να τα κάνουν όλα, πρέπει να, ε, πραγματικά να κατακαιρματιστούν έτσι ώστε να είναι καλές και επαγγελματικά, σε περίοδο κρίσης μάλιστα και στην οικογένεια. Πραγματικά το βλέπουμε. Το βλέπουμε σήμερα. Σήμερα μιλάμε για αυτό το, για αυτό το θέμα, μιλάμε για ανεργία και πιστεύω πως ως Ευρωπαϊκή, ε, πρέπει να πιέσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να βρεθεί λύση, να βρεθούν λύσεις, διαφορετικές λύσεις, άλλες για τις γυναίκες, άλλες για τους άνδρες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε την κρίση δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά για τους άντρες και για τις γυναίκες, διότι οι συνθήκες είναι διαφορετικές για τους μεν και διαφορετικές για τους δε. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να βρούμε συγκεκριμένες στοχευμένες λύσεις, διότι φυσικά και αληθεύουν όσα υπόθηκαν μέχρι τώρα, όμως... Χρειάζεται βελτίωση. Όπω είπα, χρειάζονται λύσει. Και φυσικά είναι ρητορικό το ερώτημα. Ναι, έχουμε βρει κάποια λύση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και με αυτό το ερώτημα ολοκληρώνω και θα ήθελα να πω ότι δυστυχώς δεν ε, έχει βρεθεί μια λύση αλλά δεν έχει καμία σύνδεση προς το παρόν με την ανεργία. και έχει να κάνει με το πώς πηγαίνουν να ψηφίσουν σε εκλογές οι γυναίκες και οι άνδρες, με την εκπροσώπηση των γυναικών στις, ε, στα διοικητικά συμβούλια, όπως ε, ε Όπω έχει προτείνει και η Επίτροπος Ρέντινγκ αυτή την ρύθμιση, είναι κάτι πρέπει να συζητήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Το πρώτο που θα ήθελα να σας πω είναι ότι η Πέρση δεν είναι από την εποχή του Ηρώδη. Στη Γαλλία το Μάρτιο έγινε μια ευρύτατη μελέτη και ποιο ήταν το ερώτημα, δημοσκόπηση μάλλον. Πιστεύετε ότι εν περίοδο κρίσης ε, θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα οι άντρες για την αγορά εργασίας. 63% ε, ε, των ερωτηθέντων απίτησαν καταφατικά μιλώντας για στερεότυπα. Ε, ότι ε, ο μισθός δηλαδή και η δουλειά των γυναικών είναι ad hoc ε, φαινόμενο και ότι το βασικό που πρέπει να κατοχυρώνεται είναι ο μισθός και η δουλειά των αντρών. Αυτό σημαίνει και ας με διορθώσει η Ρομπέρτα γιατί ασχολείται επισταμένα με αυτά τα ζητήματα εγώ πιστεύω ότι μιλώντας για την συμφιλίωση οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής θεωρώ διότι παραθέσατε κι εσείς ε, ε, στοιχεία για τη συμμετοχή των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια. Πιστεύω λοιπόν ότι ε, ο ίσος επιμερισμός καθηκόντων ανάμεσα στα δύο φύλλα για τις οικογενειακές ευθύνες είναι κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία. Εξάλλου από αυτού θα ήθελα να σας πω πως οι γυναίκες δεν είναι λογικές από συναισθηματικής τουλάχιστον πλευράς αφαιρούν από τους άντρες ε, τη χαρά του να μετάσχουν στην ανατροφή ε, των παιδιών. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να βρούμε μια νέα ισορροπία και όλοι πρέπει να ε, συνεργαστούμε και τα δύο φύλλα για να μπορέσουμε να βρούμε αυτή τη νέα ισορροπία. Η κυρία Σάμεκ μήπως θέλει να κάνει ένα τελευταίο σχόλιο πριν περάσουμε στον επόμενο γύρο. Ναι, κατά την άποψή μου το πρόβλημα είναι να μπορεί κανείς να επιλέξει Συνεπώς να υπάρχει μια προσφορά υπηρεσιών που επιτρέπουν την επιλογή. Πράγματι υπάρχει πρόβλημα επιμερισμού των ρόλων εντός της οικογένειας. Επ' αυτού μπορούμε να εργαστούμε μέσω παρεμβάσεων, ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης, κατάρτισης κλπ από την πολύ μικρή ηλικία. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα όμως είναι η έλλειψη υπηρεσιών, προσφοράς υπηρεσιών περίθαψης θεραπείας που επιτρέπουν τελικά την ε, επιλογή να μπορεί να δουλέψει κανείς έχοντας παιδιά. Το πρόβλημα είναι ότι με αυτή την κρίση, με τις περικοπές όσον αφορά τις δημόσιες δαπάνες, όλες αυτές οι περικοπές ε, ε, έχουν το κίνδυνο να μειωθούν και οι δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών υπηρεσίας, περίθαλψης, θεραπείας, περισσότερο από τις άλλες δαπάνες. Υπάρχει και ένα πρόβλημα προτεραιοτήτων όσον αφορά τις επιλογές των οικονομικών πολιτικών. Η περικοπή των δημοσίων δαπανών για τις υπηρεσίες αυτές φροντίδας, άρα τελικά η φροντίδα θα πέσει πλάτη των γυναικών, άρα θα μειωθεί περισσότερο η απασχόληση των γυναικών διότι οι γυναίκες ασχολούνται με αυτές τις υπηρεσίες κατά πολύ. Πράγματι αληθεύει, υπάρχει πρόβλημα νοοτροπίας, στερεοτύπων, αλλά υπάρχει και ένα πρόβλημα πολιτικών ε, και της παροχής των υπηρεσιών. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώνουμε τώρα τον πρώτο γύρο και περνάμε στο δεύτερο. Θα κάνουμε κάποιες τροποποιήσεις εδώ στο πάνελ. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε λοιπόν. Η κυρία Στάρκ μπορεί να αρχίσει, έχει και μια παρουσίαση. Και οι υπόλοιποι παρακαλώ ελάτε μαζί μας, καθίστε κοντά μας. Κύριε Μονινουέβο, και καθώς περιμένουμε να ετοιμαστούν όλα, θα ήθελα να κάνω μία μικρή ανακοίνωση. Έχουμε δύο ομάδες επισκεπτών σήμερα μαζί μας αν δεν κάνω λάθος, η πρώτη ομάδα από ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Γερμανία και ε, δεύτερη ομάδα από τη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης. Χαίρομαι πολύ που ήρθατε σήμερα. Όπως σας είπα, προχωράμε τώρα στο δεύτερο πάνελ, αναλύσεις των διάφορων έμφυλων απόψεων στην αγορά εργασίας που έχουν σχέση με την απασχολησιμότητα ανδρών και γυναικών. Πρώτη θα μιλήσει η κυρία Αγνιέτα Στάρκ, θα μιλήσει για τις επιπτώσεις των ε, εκπαιδευτικών επιδόσεων στην απασχολησιμότητα. Έχουν οι νέες γυναίκες πλεονέκτημα σε σχέση με τους νέους άνδρες. Είναι επίτιμη καθηγήτρια, έχει δημοσιεύσει πάρα πολλά επιστημονικά βιβλία. Έχω διαβάσει και μερικά από αυτά και μπορώ να πω ότι είναι πάρα πολύ καλά. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα είναι οικονομική θεωρία, λογιστική θεωρία, οικονομική αλλαγή οι διεθνείς συγκρίσεις της ε, έμιστης και άμυστης εργασίας. Παρακαλώ, κυρία Στάρκα, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Η συζήτηση για την ισότητα των φύλων πολλές φορές έχει την τάση να είναι καταθλιπτική. Χαίρομαι λοιπόν πάρα πολύ που μπορώ να αρχίσω να μιλώ για τις επιτυχίες των τελευταίων 15 ετών. Επιτυχίες ε, δηλαδή η αύξηση Τη πρόσβασης των γυναικών στην εκπαίδευση. Ήταν πραγματικά εκπληκτική η πρόοδο. Οι γυναίκες έχουν αγωνιστεί σκληρά και συνέχεια για να μπορούν να συμμετέχουν σε όλα τα επίπεδα της ε, εκπαίδευσης. Και πραγματικά μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα, τα θετικά αποτελέσματα παντού στον κόσμο. Η εκπαίδευση των γυναικών σήμερα θεωρείται ένα ένας παράγοντας κλειδί για την οικονομική και δημοκρατική ανάπτυξη των χωρών. Και θα σας δώσω ορισμένα παραδείγματα σε λίγο. Σήμερα οι γυναίκες συμμετέχουν και με επιτυχία μάλιστα σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλέ φορές έχουν καλύτερες επιδόσεις από τους άνδρες και τα αγόρια, τα οποία τώρα τείνουν να παραμελούν ορισμένες ευκαιρίες που τους παρέχονται για εκπαίδευση. Και αυτό είναι κάτι καινούριο. Αυτό δεν ίσχυε πριν από κάποια χρόνια. Ε, υπάρχουν εκθέσεις του ΟΣΑ και όπως ξέρετε ο ΩΣΑ είναι μεγαλύτερος από την Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 κρατών μελών και σύμφωνα λοιπόν με δεδομένα του ΩΣΑ τα αγόρια έχουν μεγαλύτερη τάση να εγκαταλείψουν το σχολείο χωρίς επιτυχίο. Και αν δείτε αυτή εδώ τη διαφάνεια, θα δείτε για τους... Ε, θα δείτε 11,3% των γυναικών και 15,3% των ανδρών εγκαταλείπουν το σχολείο πριν ολοκληρωθεί η δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Είναι ρεκόρ αυτό που έχουν. Το αρνητικότατο ρετό, ρεκόρ παρατηρείται στην Ισπανία, όπου 30% των νέων ανδρών εγκαταλείπουν προώρα το σχολείο και 22% των γέων γυναικών. Η χώρα με τα χαμηλότερα ποσοστά είναι η Τσεχία και η Σλοβακία. Μόνο 5,4% των ανδρών εγκαταλείπουν προώρα το σχολείο και στη Σλοβενία επίσης με 2,5% των γυναικών που εγκαταλείπουν το σχολείο προτού ολοκληρώσουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Πριν πάρουν απολυτήριο ηλικίου δηλαδή. Δεν είναι λοιπόν ζήτημα βιολογίας αυτό, διότι τα νούμερα έχουν αλλάξει. Ήταν διαφορετικά 30 χρόνια πριν. Και φαίνεται ότι δεν φταίει κατά ανάγκη η αγορά εργασία όμω, αλλά το ζήτημα είναι πολύ πιο περίπλοκο και είναι ένα συνδυασμός, ένα πλέγμα ζητημάτων. Και πλέον το απολυτήριο δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι απαραίτητη προπόθεση για να μπει κανεί στην αγορά εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πρέπει να, πραγματικά να αποτρέψουμε του νέου ανθρώπου από το να εγκαταλείψουν πρόωρα το σχολείο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Οι νέε γυναίκε τώρα είναι πολύ περισσότερο πιθανέ να ολοκληρώσουν το, δευτεροβάθμια εκπαίδευση από του άντρε, αλλά επίση και να πάρουν πτυχίο τρίτο βάθμιας εκπαίδευσης. Κοιτάξτε τώρα αυτό το διάγραμμα. Δεν είναι και πολύ ωραίο διάγραμμα, αλλά κοιτάξτε τις ε, πράσινε μπάρε. Πράσινες μπάρες λοιπόν δείχνουν τις ε, επιδόσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ανάλογα με το φύλλο στην Ευρώπη των 27 κρατών μελών. Από ηλικίες 30 έως 34 μόνο γυναίκες. Το ανώτατο λοιπόν, ε, η ανώτατη τιμή είναι 60% και μετά 55% και θα δείτε ότι υπάρχει ένα μεγάλο φάσμα χωρών που βρίσκονται γύρω στο 50%. 50% δηλαδή γυναικών 30 έως 34, 34 ετών δεν έχουν πάρει το επιτυχία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ε, εκεί που βλέπετε χ δεν σημαίνει ότι έχουν χαμηλά ποσοστά, σημαίνει ότι δεν είχαμε δεδομένα. Τώρα, ας περάσουμε στους άντρες, στην επόμενη διαφάνεια. Εδώ βλέπετε στο διάγραμμα ότι ούτε μία χώρα δεν φτάνει το 50%. Υπάρχουν ε, χαμηλότερα ποσοστά. Συγκεντρώνεται ο μέσος όρος γύρω στο 40% το οποίο είναι και μάλιστα ιδιαίτερα χαμηλό και μάλιστα πολύ χαμηλότερο για κάποιες άλλες χώρες και αυτές είναι κάποιες αλλαγές που έχουν παρατηρηθεί τα τελευταία 40 χρόνια, οι οποίες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Τι βλέπουμε λοιπόν. Βλέπουμε ότι οι γυναίκες προχωράνε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αλλά επίσης έχουν να αντιμετωπίσουν εκτός από όλες τις άλλες δυσκολίες και ταξικές διαφορές. Αν δείτε τους αποφύτους πανεπιστημίου, των οποίων οι γονείς δεν είχαν πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τότε θα δείτε ότι και πάλι οι γυναίκες υπερέχουν πάνω από το 10% των γυναικών ε, με γονεί που δεν έχουν παρελθόν τρίτο βάθμας εκπαίδευσης παίρνουν πτυχίο σε σχέση με τους άνδρες και η Ελλάδα, η Ισλανδία, η Σλοβακία και η Ισπανία είναι από τις χώρες με τα μεγαλύτερα αυτά ποσοστά γυναικών πτυχιούχων. Υπάρχουν, ό, βλέπετε, δυσκολίες τι οποίες όμως έχουν ξεπεράσει οι γυναίκε, έχουν δείξει επιτυχία. Τώρα, σε κάθε επίπεδο εκπαίδευση, υπάρχει κίνδυνος ανεργίας. Ο κίνδυνο όμως αυτός μειώνεται όσο αυξάνεται το επίπεδο εκπαίδευση. Αυτή η κρίση που συνεχίζεται έχει χτυπήσει, έχει πλήξει περισσότερο τους ανθρώπους που δεν έχουν καν πτυχίο ε, απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Και οι άντρες έχουν πληγεί πολύ περισσότερο από ό,τι οι γυναίκες. Ίσως ενδεχομένως επειδή έχουν εξαφανιστεί ορισμένα επαγγέλματα που θεωρούνταν παραδοσιακά αντρικά, δηλαδή στις, ε, στις, στον κατασκευαστικό κλάδο. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι οι γυναίκες δεν είχαν προβλήματα. Το ζήτημα της ισότητας είναι ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να έχουν προβλήματα. Μπορεί να μην είναι τα παραδοσιακά προβλήματα που είχαν στο παρελθόν, εξακολουθούν όμως να υπάρχουν ιδιαίτερα αυξημένα προβλήματα. Ας δούμε τι συμβαίνει όταν βρίσκεσαι στην αγορά εργασίας. Εδώ το επίπεδο μόρφωση παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στι απολαυέ σου. Υψηλότερο επίπεδο μόρφωση σημαίνει χαμηλότερο κίνδυνο ανεργία και Υψηλότερο επίπεδο μόρφωσης γενικότερα σημαίνει καλύτερος μισθός. Όμως, σε όλους τους τομείς της αγοράς εργασίας, οι άνδρες υπερέχουν σε νούμερα απέναντι στις γυναίκες και μιλάμε πάντα για ανθρώπους που έχουν τα ίδια προσόντα. Τώρα, αν πάμε στην τρίτο βάθμια εκπαίδευση οι γυναίκες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ε, ε, οι γυναίκες δεν αποκομίζουν τα ε, περισσότερο, περισσότερα ωφέλη, χρηματικά ωφέλη, έχοντα επιτυχία τριτοβάθμια εκπαίδευση. Γιατί λοιπόν το κάνουν. Είναι, υπάρχει κάτι ενδιαφέρον που έχουμε παρατηρήσει. Υπάρχει μειωμένο ενδιαφέρον στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από τους άνδρες παρά το γεγονός ότι με το πτυχίο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κερδίζουν περισσότερα δεν είναι οικονομικά λογικό, σωστά. Επίσης, οι γυναίκες θεωρούνται ότι δεν ε, είναι ικανές να πάρουν οικονομικά λογικές αποφάσεις. Όμως με αυτό που μόλις είπα φαίνεται πως ε, η κατάσταση αυτή σε έχει συμπεριλάβει και τους άντρες. Η εκπαίδευση δεν έχει τα ίδια στάδια ολοκλήρωση σε άνδρε και γυναίκε. Υπάρχουν άλλοι τομεί παραδοσιακά ανδρικοί και άλλοι παραδοσιακά γυναικοί στην εκπαίδευση. Ορισμένοι βέβαια έχουν ε, τονώσει τα στερεότυπα. Για παράδειγμα, το μέρος της περίθαλψης. Εάν κάποιος είναι νοσηλευτής σε μονάδα αποκλειστικής θεραπείας, η δουλειά αυτή δεν είναι μόνο χειρονακτική. Η δουλειά αυτή απαιτεί υψηλά τεχνικά και τεχνολογικά προσόντα. Απαιτεί μεγάλο ποσοστό ακρίβεια σε συνδυασμό με συμπόνια και ικανότητα επικοινωνίας. Και ένας ε, υψηλά εκπαιδευμένος και καταρτισμένος ο μηχανικός, ο οποίος είναι ο καλύτερος του τμήματός του στην μεγάλη πολυεθνική του, κατά πάσα πιθανότητα εξαρτάται πολύ, ε, περισσότερο η δουλειά του στην ε, τεχνική της επικοινωνίας από ό,τι σε άλλους τομείς. Οι ανάγκες τώρα στην εκπαίδευση και την κατάρτιση είναι ένα δύσκολο θέμα. Γνωρίζουμε τι δεν κάνουν, αλλά δεν ξέρουμε καθόλου τι συμβαίνει, ποιες είναι οι αιτίε. Είναι πολύ εύκολο να τα βάλουμε όλα σε ένα τσουβάλι και να πούμε ότι όλος ο κλάδος είναι προβληματικός, αλλά πιστεύω ότι πραγματικά αυτό που χρειάζεται είναι να μάθουμε τι γίνεται ακριβώς, ποιος συνεισφέρει, τι κάνουν οι γυναίκες για τις οικογένειές τους, ε, φροντίζουν οικογένεια, φροντίζουν καριέρε, ποιες είναι οι αποφάσεις που λαμβάνουν, παίρνουν τι σωστέ, παίρνουν τις λάθο. Είναι όμω πολύ επικίνδυνο να παίρνει μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων και να τους, ε, να τους, ε, να τους βάζεις σε αρνητική ταμπέλα. Δεν μπορούμε να υποθέσουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν κάνουν τίποτα και είναι αδρανείς. Πιστεύω πως είναι πάρα πολύ σημαντικό να μάθουμε τι ακριβώς κάνουν οι νέοι στην Ευρώπη και τι σκέφτονται. Οι ομάδες αυτές διαφέρουν πάρα πολύ από χώρα σε χώρα. Έχουν τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Η Eurofound έχει δημοσιεύσει μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα έκθεση και σας καλώ να την διαβάσετε. Δεν θα πω εγώ σε λεπτομέρειες, αλλά πραγματικά διαβάστε την διότι από αυτήν την έρευνα φαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα μόνο με ένα με μια ομάδα όπλων. Αν, όταν έχεις γυναίκες με υψηλά προσόντα που χρειάζονται πρόσβαση στην αγορά εργασίας, είναι κάτι τελείως διαφορετικό από όταν έχεις άνδρες με χαμηλά προσόντα που δεν μπορούν να μπουν στην αγορά εργασίας ή νέους άνδρες οι οποίοι έχουν προσόντα τα οποία όμως δεν ε, είναι πια επιθυμητά από την αγορά εργασία. Είναι τελείω διαφορετικά τα μέσα λοιπόν που χρησιμοποιούμε στην κάθε περίπτωση. Τώρα, αν δούμε τι γίνεται με την μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας, θα δούμε ότι το φύλλο παίζει καθοριστικό ρόλο. Οι νέες γυναίκες πολύ συχνά έχουν ε, προσωρινές ε, δουλειές και προσωρινές θέσεις εργασίας, αλλά έχουν όμως κάποια δουλειά. Πώς μπορούμε λοιπόν να τις βοηθήσουμε να εντάξουν αυτές τις ε, προσωρινές δουλειές στον, στο επαγγελματικό τους βιογραφικό και πώς μπορούμε να πείσουμε τους άνδρες να συνεχίσουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση όταν αυτοί δείχνουν τάση ε, απώλειας ενδιαφέροντος προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τώρα οι μετανάστες, οι νέες γυναίκες, οι νέες και οι νέοι άνδρες είναι, ε, είναι πρόβλημα. Έχει γίνει μια εις μελέτη του ΟΣΑ η οποία δείχνει ότι η γεωγραφική συγκέντρωση έχει να κάνει με τα σχολεία, με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Και πραγματικά φαίνεται από αυτό ότι η εκπαίδευση και το επίπεδο εκπαίδευση στι γυναίκε παίζει ρόλο. Οι γυναίκε αυτές θα έχουν πολύ καλύτερο μέλλον εάν διανεμηθούν περισσότερο ομαλά στα, διά, στα διάφορα ε, σχολεία, στα διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Τώρα, τι γίνεται μετά την εκπαίδευση. Μιλάμε πολλέ φορέ για το ότι οι γυναίκε έχουν υπερβολικά προσόντα. Πρέπει όμω να δούμε ότι εξίσου ανησυχητικό είναι όταν οι άνδρε δεν έχουν επαρκή προσόντα. Στη Νότια Κορέα υπάρχει πολύ μεγάλο ποσοστό ε, πτυχιούχων αποφύτων τριτοβάθμιας εκπαίδευση. Έχουν υπερβολικά προσόντα δηλαδή και αυτό είναι όντω ένα πρόβλημα. Είναι λοιπόν πάρα πολύ χρήσιμο για μας να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που έχουμε να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν αυτά που ξέρουμε, ότι δηλαδή πολλές φορές τα υψηλά προσόντα των γυναικών δεν λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από τους εργοδότες. Επίσης ότι οι εργοδότες κοιτάζουν αν γυναίκες έχουν παιδιά ή όχι και αυτό επηρεάζει τις αποφάσεις τους. Και επίσης κοιτάζοντας προς το μέλλον. προς το τι χρειάζεται να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση από το, μέχρι το 2035, μέχρι το 2040. Αυτοί οι άνθρωποι που θα χτίσουν την Ευρώπη τότε είναι αυτοί οι άνθρωποι που πηγαίνουν σχολείο τώρα, σήμερα. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να είναι είναι περίεργοι, πρέπει να είναι δημιουργικοί. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να δημιουργήσουμε μια δημιουργική καινοτόμα περίεργη γενιά. Η εκπαίδευση δεν λύνει τα πάντα, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική και η εκπαίδευση και η παιδεία δεν προορίζεται μόνο για, τον για την αγορά εργασίας, αλλά και για την διαμόρφωση της προσωπικότητας. Οι νέοι άνθρωποι προσπαθούν να συλλέξουν γνώσεις, να συγκεντρώσουν γνώσεις, να τις χρησιμοποιήσουν και πιστεύω πως η Ευρώπη αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ένα σοβαρό πρόβλημα όσον αφορά την γνώση και την εκπαίδευση. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ την Ανιέτα Στάρκ παρέμβασή σας πραγματικά μας στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα, το οποίο φάνηκε και από το βιβλίο σας, το οποίο έχω διαβάσει. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο σε εσάς για ερωτήσεις και πρώτη η Κατρίνα Νεβεντάλοβα, η οποία είναι σκιώδης εισηγήτρια στη γνωμοδότηση της Επιτροπής Γυναικών για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων γυναικών. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω στα σλοβακικά. Φορές τα ακουστικά σας παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και ζητώ συγγνώμη ταυτόχρονα διότι είχα ανηλυμένες υποχρεώσεις και έφτασα καθυστερημένα και λυπάμαι αν επαναλάβω ήδη υποθέντα. Είναι ενδιαφέρον να μιλώ μετά την προλαλήσασα, γιατί συμφωνώ με πολλά από αυτά που είπε. Είπατε ότι η εκπαίδευση δεν είναι η πανάκια, δεν είναι η λύση για τα πάντα, αλλά σίγουρα θα βοηθήσει στην επίλυση των προβλημάτων, αλλά είναι μακροχρόνια διαδικασία. Δεν θα λυθούν τα προβλήματα άμεσα, αλλά είναι το βασικό εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς και να το διαθέτει κατά τη διάρκεια της ζωής του. Είναι σημαντικό και απαραίτητο να εξακολουθήσουν οι επενδύσεις για την παιδεία και να την υποστηρίζουμε και θα είναι στον πυρήνα της παρέμβασής μου. Αν δούμε το ποσοστό ανεργίας των νέων, 23,5% ήταν το Μάρτιο, αρκετά υψηλό. Ταυτόχρονα θα πρέπει να δούμε και τα 2 εκατομμύρια που είναι θέσεις εργασίας διαθέσιμες που δεν μπορούν να καλυφθούν από τα άτομα λόγω ελλείψης προσόντων. Αυτό λοιπόν που θα πρέπει να επιλύσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι και η βάση της προτάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χάρη σοσιαλιστική ομάδα που στηρίζει αυτή την ιδέα και έγινε πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όλα αυτά λοιπόν βασίζονται στη μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος. Πρέπει να δώσουμε σημασία στην παιδεία. Θα συζητήσουμε το θέμα αυτό για να μην το συζητήσουμε το ζήτημα σε 5, 10, 15 χρόνια, γιατί πρέπει να συζητηθεί σήμερα. Είναι διθωτικό ζήτημα. Αν δούμε τους ε, άνεργους νέους που έχουμε σήμερα, θα πρέπει να λάβουμε ότι 60% των αποφύτων πανεπιστημίων είναι γυναίκες αλλά άμα δούμε την αγορά εργασίας, πού βρίσκονται αυτές οι γυναίκες. Διότι αν δούμε τις θέσεις που κατέχονται, οι άντρες είναι πιο επιτυχείς στο να βρουν δουλειά. Και αληθεύει ότι αν μια γυναίκα προσπαθεί να βρει δουλειά, ο εργοδότης πάντα τη ρωτήσει «Πότε θέλετε να κάνετε παιδιά» ε, και ο εργοδότης προτιμά έναν άντρα να προσλάβει άντρα γιατί είναι σίγουρος ότι δεν θα φύγει για κάποια χρονική περίοδο ο άντρας. Νομίζω ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε και τις νέες γυναίκες ως επιχειρηματίες. Και αυτό είναι απαραίτητο. Πρέπει να υποστηρίξουμε τις γυναίκες. Να μην φοβούνται να δημιουργήσουν δική τους επιχείρηση που θα μπορούσε να είναι αρκετά επιτυχής ούτως ώστε να παράσχει εισόδημα για εκείνη χωρίς να χρειάζεται να ανησυχεί για το αν θα έχει παιδιά ή όχι και αν κάποιος θα την απολύσει για κάτι τέτοιο. Θα είναι δική της επιχείρηση και μπορεί να την ελέγξει. Máme tu nic, čiže máme ľudí, ktorí sú mladí, nie sú ani na trhu práce, ani sa nezdelávajú, ani sa... Έχουμε νέους που όπως είπατε δεν κάνουν τίποτα, δεν σπουδάζουν, δεν εργάζονται, και είναι μια αρνητική τάση. Και πρέπει να του ενεργοποιήσουμε αυτού του νέου. Υπάρχουν πολλά προγράμματα. Η νεότη ενδράση, παραδείγματο χάρη τη Ευρωπαϊκή Ενώση, το Youth in Action, που βοηθά αυτά τα άτομα να αποκτήσουν άτυπη, όπω αποκαλείται, εκπαίδευση. Και αν δεν βρουν δουλειά, μπορούν να αποκτήσουν κάποιε δεξιότητε μέσω αυτή τη άτυπη εκπαιδεύσεω ακόμα και αν δεν είναι κλασική παιδεία. Αλλά και αυτό είναι σημαντικό μέτρο. Και άλλος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να βοηθήσουμε τις γυναίκες στην αγορά εργασίας είναι να υποστηρίξουμε κορίτσια να σπουδάσουν θέματα όπως επιστήμες, μαθηματικά, διότι στο μέλλον ίσως θα χρειαζόμαστε περισσότερους ανθρώπους που θα έχουν εκπαιδευτεί σε αυτούς τους τομείς Άρα να μην έχουμε μόνο τα αγόρια που θα σπουδάζουν μαθηματικά. Ίσως κάποια μέρα κάποια γυναίκα μπορεί να αναπτύξει κάποια νέα μαθηματική θεωρία. Αυτό όμως είναι και ένα θέμα που θα πρέπει να επιληθεί στο δημοτικό ή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Θα πρέπει οι δάσκαλοι να στηρίξουν τα κορίτσια να διαλέξουν τα θέματα. Κοιτάζω προ τον πρόεδρο, καταλαβαίνω θέλει να μα σταματήσει. Θα πάω όσο πιο γρήγορα γίνεται για να τελειώνω. Τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να βοηθήσουμε τι γυναίκε να μπορούν να συμφιλιώσουν επαγγελματική και οικογενειακή ζωή. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να παράσχουμε πρόνοια για τα παιδιά. Αν αποφασίσει λοιπόν μια γυναίκα ότι θα αποκτήσει παιδί, να έχει κάπου που να μπορεί να ξέρει ότι θα προσέξουν το παιδί της και θα πρέπει το κράτος να εγγυάται κάτι τέτοιο. Διότι γνωρίζουμε ότι αυτή η γυναίκα πρέπει να είναι σίγουρη ότι όταν θα επιστρέψει μετά την άδεια τη γονική θα πρέπει να πληρώνεται με τα ίδια χρήματα και όχι 12% λιγότερο όπως ισχύει τώρα. Υπάρχει διαφορά αμοιβή μεταξύ των δύο φύλων Έχω περίπου τέσσερι σελίδε με προτάσεις και θα σταματήσω γιατί υποβάλλω. Ευχαριστώ την προσοχή σα. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Χαίρομαι πολύ που έχετε τέσσερι σελίδε. να μας δώσετε. Με τα χαράς να τι δούμε. Δυστυχώ πρέπει να προχωρήσουμε όμω. Η κυρία Ζούμπερ έχει το λόγο τώρα. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ζητήσω συγγνώμη γιατί είχε προβλεφθεί να είμαι στο επόμενο πάνελ αλλά λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν είναι δυνατό αυτό. Θα ήθελα παρόλα αυτά να κάνω ε, κάποια σχόλια για το υποσυζήτηση θέμα. Δηλαδή η σχέση της εκπαίδευσης με την απασχολησιμότητα και την αγο... θέση στην αγορά εργασίας. Θα ήθελα να καταθέσω κάποιες σκέψεις εντάχει. Σε διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων και δική μου, αυτό που συμβαίνει είναι πως ένα μεγάλο ε, τμήμα των νέων με τις περισσότερες δεξιότητες δεν βρίσκουν δουλειά στη χώρα τους. Είναι μια πραγματικότητα που αληθεύει λένε ένα και περισσότερο. Οι που έχουν τις υψηλότερες δεξιότητες ή δεν απασχολούνται ή οι εργασιακές τους ε, συνθήκες θα χαρακτηρίζονταν ε, επισφαλείς και σαφίστατα χειρότερες από αυτές που ισχύουν σε άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, εγκαταλείπουν το εκπαιδευτικό σύστημα, διότι βλέπουν ότι δεν, θα, δεν θέλουν να ζουν με τις υποτροφίες αυτοί που έχουν τα μάστερ, τα διδακτορικά. Χρειάζονται μια πραγματική πάγια θέση απασχόλησης. Ε, τροφοδοτείται ένα μοντέλο χαμηλών μισθών Ε, εξαιτίας του οποίου κάποιοι ε, προτιμούν ε, να παραμείνουν στην αγορά εργασίας, άλλοι πάλι όχι. Από οικονομικής πλευράς είναι σοβαρές οι συνέπειες, αλλά σίγουρα δημιουργεί μείζωνα προβλήματα στη χώρα, διότι πολλοί νέοι εγκαταλείπουν τη χώρα ενώ έχουν γίνει επενδύσεις από πλευράς του κράτους για την εκπαίδευσή τους. Και πολλές φορές, και γνωρίζω προσωπικά διάφορες περιπτώσεις, χρειάζεται ο υποψήφιος να παραλείψει, να μην συμπεριλάβει τις δεξιότητες του στο βιογραφικό του σημείωμα, γιατί έχει υπερβολικές ε, δεξιότητες για τις λιγοστές ευκαιρίες που υπάρχουν πλέον στην Πορτογαλία για να βρει κάποιος δουλειά. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Υπάρχει και μια άλλη τάση στην οποία θα ήθελα να αναφερθώ. Ένας φοιτητής σήμερα γνωρίζοντας την πραγματικότητα, δεν έχει κανένα σοβαρό κίνητρο για να συνεχίσει την εκπαίδευσή του, διότι ε, ένας φίλος, ένας γνωστός που είναι 10 χρόνια μεγαλύτερος και έχει ε, ολοκληρώσει έναν ανώτερο κύκλο σπουδών, είναι άνεργος. Δεν βλέπει λοιπόν για ποιο λόγο πρέπει να συνεχίσει να φυτά στο πανεπιστήμιο. Δεν κρίνει ότι ε, θα έχει καλύτερες ευκαιρίες στατιστικώς, πως ξέρουμε ότι αυτό δεν επαληθεύεται γνωρίζουμε ότι το επίπεδο της εκπαίδευσης σε σχέση με τις δυνατότητες της εξέβρεσης θέσης εργασίας δείχνει ότι κάποιος που έχει υψηλότερες δεξιότητες έχει περισσότερες πιθανότητες ε, να βρει μια θέση απασχόλησης. Βλέπουμε λοιπόν μια κατάτμιση της αγοράς εργασίας και μεγάλες ε, διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Ε, το ζήτημα είναι να δούμε ποιες διαρθρωτικές πολιτικές έχουν δημιουργήσει ποιες καταστάσεις στην αγορά εργασίας ε, των κρατών μελών για να καταλάβουμε πού πρέπει να γίνουν οι προσαρμογές. Ε, αυτό που χρειάζεται είναι μεγαλύτερες δημόσιες επενδύσεις για να διορθωθούν αυτές οι διαρθρωτικές αλλαγές, Πρόεδρο. Σας ευχαριστώ. Κυρία Στάρκ, μήπως θα θέλατε να απαντήσετε σε αυτά τα δύο σχόλια. Ναι. Ε, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναλύσουμε εις βάθος ακριβώς τα προβλήματα που προσπαθείτε να λύσετε και να εξετάσετε κάθε επιμέρους περίπτωση, διότι στις περισσότερες χώρες ε, της Ένωσης ε, υπάρχει το πρόβλημα το να βρεθούν στις κατάλληλες θέσεις αυτοί που έχουν υψηλή δεξιότητα. Σε άλλες χώρες πάλι αυτοί που έχουν υψηλές δεξιότητες δεν μπορούν να βρουν την κατάλληλη θέση εργασίας. Ε, δεν υπάρχει αντιστοίχηση και ξέρουμε επίσης ότι και ο ευρωπαϊκός πληθυσμός και γνωρίζουμε επίσης ότι χρειαζόμαστε το ταλέντο και αυτές τις δεξιότητες για να βρούμε μία λύση. Αλλά δεν είναι εύκολο επίλυτο αυτό το πρόβλημα και αναφερθεί στις χώρες ε, όπου υπάρχουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Υπάρχει μια ολόκληρη γενιά ανθρώπων ε, με υψηλές δεξιότητες ή υψηλέ ειδικευμένων εργατών που ε, αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Πώς μπορούμε να του επανακαταρτήσουμε, να του επαναπροσανατολίσουμε να βρούμε τρόπους επίσης ε, οι νέοι να ε, κατευθυνθούν προς μια ε, κατάλληλη επαγγελματική σταδιοδρομία. Γι' αυτό δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα ενιαίο μοντέλο, δεν μπορεί να λειτουργήσει μια τέτοια λύση. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κυρία Στάρκ. Θα συνεχίσουμε με το πρόγραμμά μας τώρα. Θα ήθελα να καλέσω τους επόμενους ομιλητές. Ο κύριος Ντάνιελ Μόλιβουέδα από το Eurofound που θα μας παρουσιάσει την ε, κατάσταση των ε, νέων στην αγορά εργασίας ε, μιλώντας συγκεκριμένα για τα αποτελέσματα που έχουν τα συστήματα περίθελψης των παιδιών και άλλων εξαρτωμένων μελών της οικογένειας στις επαγγελματικές επιλογές του καθενός και στην κατάσταση της αγοράς εργασίας για τους νέους. Ε, από το 2010 είσαστε στο Eurofound. Προ αυτού είχατε εργαστεί σε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο παροχής κοινωνικών υπηρεσιών όπου ασχοληθήκατε με τις πολιτικές για ε, τα παιδιά, ή για την οικογένειες, για την πνευματική υγεία. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κάναμε λοιπόν μία μελέτη για το εργαστήριο. Αυτό εξετάσαμε τρία στοιχεία όσον αφορά την κατάσταση που επικρατεί για τους ε, νέους με, που ασκούνται με τη φροντίδα στην αγορά εργασίας. Κάναμε και δευτερογενή ε, ανάλυση των δικών μας ε, ερευνών και του Ευρωβαρομέτρου 76,2 και την επισκόπηση του εργατικού δυναμικού να δούμε ποια είναι η κατάσταση στην αγορά εργασίας όσον αφορά τους νέους που έχουν παιδιά, ή που φροντίζουν ηλικιωμένους συγγενείς. Εξετάσαμε και τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ εκείνων που παρέχουν φροντίδα στο σπίτι και σε σχέση με τους νέους στην αγορά εργασία εστιαζόμενοι επί των γυναικών που τείνουν όπως γνωρίζουμε να είναι εκείνες που αναλαμβάνουν αυτές τις φροντίδες στο σπίτι και συμπεριλάβαμε με σύντομη περιγραφή κόστους, ανάλυση κόστους-οφέλους και των οικονομικών ωφελών επενδύσεων ε, τέτοιων ε, υπηρεσιών περίθαψη και φροντίδα στην Αυστρία. Όσον αφορά τώρα του νέου που φροντίζουν ηλικιωμένου συγγενεί, αυτό που ανέφερα, έχουμε κάποια στοιχεία από το Ευρωβαρόμετρο που δείχνει ότι εν γέννη στην Ευρώπη, δείχνουν αυτά τα στοιχεία, 2,2 εκατομμύρια άνθρωποι είναι μεταξύ της ηλικίας 15 με 30 ετών και φροντίζουν ηλικιωμένο συγγενείς είναι εξίσου δραστήριοι και ανενεργοί. Ξέρουμε ότι οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να αναλάβουν φροντίδα ηλικιωμένου στο σπίτι και από το ευρωβαρόμετρο βλέπουμε ενδιαφέρον ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των φύλων όσον αφορά την φροντίδα πλήρους απασχόλησης και μερικής απασχόλησης. Σε πλήρη απασχόληση ένα μισή εκατομμύριο γυναίκες ασχολούνται με την πλήρη φροντίδα ηλικιωμένων έναντι 700.000 ανδρών, δύο φορέ περισσότερε γυναίκε από άντρε. Όσον αφορά τη μερική απασχόληση, όσον αφορά τη φροντίδα ηλικιωμένων, υπάρχει καλύτερη ισορροπία μεταξύ των φίλων. 500.000 γυναίκε, 500.000 άντρε φροντίζουν ηλικιωμένου στο σπίτι. Επιπλέον πρέπει να τονίσουμε την ασταθή κατάσταση που επικρατεί όσον αφορά τους ανθρώπους στην αγορά εργασίας φαίνεται να θεωρούν ότι είναι πολύ πιο πιθανό να χάσουν τη δουλειά τους λόγω της κρίσης και είναι πιο απεσιόδοξοι για τη δυνατότητα να βρουν μια νέα δουλειά αν χάσουν την παρούσα δουλειά τους και τείνουν να αλλάζουν δουλειές και εργοδότες πιο συχνά από εκείνους που ποτέ δεν έπρεπε να φροντίσουν ηλικιωμένο συγγενή. Αυτό ήδη μας δείχνει κάποιες τάσει. κυρίως αν κάποιος φρόντιζε ηλικιωμένο κατά παρελθόν. 15% ανθρώπων κάτω από το 30. Κάτω από 30 ετών αλλάζουν τουλάχιστον 5 δουλειέ. Δεν είναι πολύ σταθερή η κατάστασή του στην αγορά εργασία. Αυτά είναι τα στοιχεία για ανθρώπους που φροντίζουν ηλικιωμένο συγγενή όσον αφορά τους νέους Νέους τι εννοώ. Γονείς από 18 μέχρι 29. Τέσσερα στοιχεία να προσέξουμε. Μεγάλος αριθμός υπάρχει νέων με παιδιά που είναι αδρανείς, ανενεργοί και θέλουν να... θα ήθελα να βρουν δουλειά αν μπορούσαν να επιλέξουν το ράριο εργασίας ελεύθερα. 80% από εκείνους που δεν είναι δραστηριοποιημένοι θέλουν αυτόν. Αν ρωτήσει κάποιου από αυτού που εργάζονται ήδη αν θέλουν να δουλέψουν περισσότερε λιγότερες λιγότερε ώρε, περισσότεροι λένε προτιμώ να δουλέψω λιγότερε ώρε. Αλλά 18% των νέων γονέων θα ήθελαν να δουλεύουν περισσότερες ώρες. Ε, στην έρευνα για την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη ε, ε, ερευνούμε την όλη κατάσταση μέσω τριών ερωτήσεων. Πόσο συχνά γύρισαν πολύ κουρασμένοι για να κάνουν τα οικογενειακά του, να ασκήσουν τα οικογενειακά του καθήκοντα, ήταν η πρώτη ερώτηση. Ε, διότι δουλειά που έκανα πολλή δουλειά στο γραφείο του. Δεύτερον, πόσο δύσκολο είναι να ανταποκριθούν στα οικογενειακά του καθήκοντα λόγω των εργασιακών του καθηκόντων δεν εξετάζουμε το πώς επηρεάζει η δουλειά τα οικογενειακό καθήκοντα, αλλά και το αντίστροφο. Τους ρωτάμε πόσο συχνά είναι δύσκολο να συγκεντρωθούν στη δουλειά τους, διότι τους απασχολούν τα καθήκοντά τους στο σπίτι. Βλέπουμε αν υπάρχει σύγκρουση εργασιακής ζωής και έχουμε ετοιμάσει δίκτυ που δείχνει τη σύγκρουση μεταξύ των δύο ζωών. Εκείνοι που έχουν φροντίσουν μικρά παιδιά είναι δύο φωσιοποιοί πιθανόν να πούν ότι έχουν προβλήματα και στο σπίτι και στη δουλειά από ότι εκείνοι που δεν έχουν παιδιά. Και τα ποσοστά είναι 20% νέων γυναικών και ανδρών με παιδιά που λένε ότι έχουν προβλήματα και στο σπίτι και στη δουλειά έναντι 10% μόνο ανδρών και γυναικών που δεν έχουν παιδιά και που αναφέρουν ότι έχουν προβλήματα. Και τέλος, όσον αφορά και φροντίζουν ηλικιωμένους συγγενείς, οι νέοι που πρέπει να φροντίσουν παιδιά ε, αισθάνονται πιο ασφα... ανασφαλείς όσον αφορά τη θέση στην αγορά εργασίας. Θεωρούν ότι είναι λιγότερο σταθερή η δουλειά τους. Η φροντίδα των παιδιών θα βοηθούσε να μειωθεί η ανισορροπία μεταξύ εργασιακής ζωής και οικογενειακής ζωής. Δουλεύουν λιγότερο ή δεν δουλεύουν καθόλου θέληση για την ποιότητα της ζωής είναι μια έρευνα που δίνει στοιχεία για τα ζητήματα που ε, αντιμετωπίζουν οι νέοι γονείς όταν προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες. Έχουμε ένα ερώτημα. Ποιες από τις μεταβλητές αντιμετωπίσατε όταν προσπαθήσατε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μέρημνας για τα παιδιά. Οι περισσότεροι νέοι με παιδιά είπαν ότι προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν 79% προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες και από αυτούς είπαν ο μεγαλύτερος φραγμός για τη χρήση των υπηρεσιών ήταν το κόστος της ε, τα παιδιά. 62% και άλλοι είπαν ότι δεν μπορούν να εξασφαλίσουν μια θέση ε, στα κέντρα φροντίδας παιδιών. Μετά ήταν η απόσταση και προβλήματα φυσικής πρόσβασης και τέλος η ποιότητα της ε, φροντίδας είναι λιγότερο ζήτημα από τα προαναφερθέντα στοιχεία. Αυτή είναι η κατάσταση λοιπόν που επικρατεί όσον αφορά τους νέους άνδρες και γυναίκες που έχουν καθήκοντα φροντίδα στο σπίτι. Ποια η σχέση όμως μεταξύ πρόσβασης σε φροντίδα για τα παιδιά και θέσεις των νέων στην αγορά εργασίας. Να προσέξουμε το ίδιο και το εδώ. Υποθέτουμε συχνά ότι αν κάποιοι έχουν παιδιά και δεν μπορούν να έχουν φροντίδα για τα παιδιά, δεν θα μπορούν να μπουν στην αγορά εργασίας. Αυτό υποθέτουμε. Από τα στοιχεία όμως του Ευρωβαρομέτρου είδαμε ότι το να μην μπουν, να μην βρουν θέση στην αγορά εργασία και να φροντίζουν ε, κάποιον συγγενή ε, στο σπίτι ε, είναι κάτι που αφορά εκείνους που ούτως ή άλλως δεν θα βρίσκαν θέση ε, ε, εργασίας. Αυτοί που έχουν λιγότερα προσόντα είναι πιθανότερο να φροντίσουν κάποιο ηλικιωμένο στενή θα βρίσκαν δουλειά ούτως ή άλλως. Και ο ΑΣΑ έχει αντίστροφο αίτιο και αιτιατό. Μεταξύ του υψηλού ποσοστού γυναικής συμμετοχής στην αγορά εργασίας και τη θεσιμότητα των φροντίδων για τα παιδιά. Υποθέτουμε κανονικά ότι αν υπάρχει καλύτερη υπηρεσία τη φροντίδα των παιδιών θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασία. Όμω τα στοιχεία δείχνουν ότι στην περίπτωση τη Δανία το αντίστροφο συνέβαινε. Όταν μιλάμε για τη σχέση μεταξύ περίθαλψη για τα παιδιά και το κόστο και τα κίνητρα από την άλλη για την ίσον αγορά εργασία, θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη όχι μόνο την τιμή τη χρήση υπηρεσιών για τα παιδιά, αλλά και τα ωφέλη και τις φορολογικές ελαφρύνσεις που χάνονται όταν μπει στην αγορά εργασίας. Όταν γίνονται μεταρρυθμίσεις του κράτους προνοίας και των φόρων θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη ότι σε κάποιες περιπτώσεις αυτές οι μεταρρυθμίσεις έχουν αντίκτυπο, σαν αντίκτυπο τη διεύρυνση του χάσματος μεταξύ των ε, φύλων, των αμοιβών των φύλων. Διότι τα ποσοστά φορολόγησης του δευτεροβάθμιου τομέα ε, είναι πιο υψηλά. Είδαμε μεταρρυθμίσεις στην Αυστραλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και στη ΣΥΠΑ και είδαμε ότι οδηγηθήκαμε σε νέο είδους διάκριση και τέλος, πιο σημαντικό να προσέξουμε ότι η επένδυση περισσότερων χρημάτων στις, ε, στη φροντίδα των παιδιών δεν είναι επανάκια όσον αφορά την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας. Σε χώρες όπως Σουηδία, η Νορβηγία, όπου υπάρχει πληρέστατο σύστημα περίθαυσης παιδιών που είναι φθηνό, έδειξαν οι μελέτες ότι περαιτέρω επενδύσεις στη φροντίδα των παιδιών δεν κάνουν μεγάλη διαφορά όσον αφορά τις, ε, την απόφαση των γυναικών να μπουν στην αγορά εργασία ή να μην μπουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις όταν ήδη υπάρχει ανεπτυγμένο σύστημα φροντίδας των παιδιών είναι σημαντικό να εστιαζόμεθα επιθεμάτων όπως είναι οι βέλτιστες συνθήκες εργασίας και πιο γενναιόδωρα συστήματα αγωνικών αδειών. Όλα αυτά καλά και άγια, αλλά σε περιόδους λιτότητας πώς μπορούμε να δικαιολογήσουμε περαιτέρω επενδύσεις στις υπηρεσίες φροντίδας παιδιών. Το επιμελητήριο εργασίας της Αυστρίας εξετίμησε το κόστος για τις υπηρεσίες περίθαλψης παιδιών ετησίως Υπολογίστηκαν τα θέματα δημιουργήθηκαν απασχόληση, ε, εκμάθηση και κέρδη για τον ε, προπολογισμό, τον κρατικό από τι επενδύσεις που γίνονται. Έγινε ανάλυση κόστο ωφέλους δηλαδή. Αυτέ είναι οι μεταβλητές που συμπεριλαμβάνονται στο κόστος, προσωπικό κόστος. Η κατασκευή νέων εγκαταστάσεων, η κατάρτιση, η χρηματοδότηση. Και όσον αφορά τα αποτελέσματα, ε, τα κέντρα φροντίδας για τα παιδιά και την έμεση απασχόληση που δημιουργείται, απασχόληση που δημιουργείται στις οικοδομές κλπ. Και τι αντίκτυπο έχει για καλύτερη συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και άλλα θέματα που είναι πιο περίπλοκο όπως η, να υπολογιστούν αύξηση κατανάλωσης. Συναρτήσει όλων αυτών υπολόγισαν τις αποδόσεις υπό τη μορφή συνεισφορών και φόρων από άμεσες και έμεσες διαδράσεις. Υπολογίζουν λοιπόν ότι έχουν τρία κέρδη βάσει των εκτιμήσεων που έγιναν. Αισιόδοξε, απεσιόδοξε, προσπαθώντας να υπολογίσουν τον αντίκτυπο των συμπροματικών κέντρων περίθαλψης παιδιών. Δηλαδή πόσες περισσότερες γυναίκες θα μπορούν να δουλέψουν. έχουμε τρία ενδεχόμενα. Ακόμα και στο επεσιόδοξο βλέπουμε ότι η επένδυση σε κέντρα περίθαψης παιδιών μετά από τέσσερα χρόνια αποπληρώνει την επένδυση. Διότι βλέπετε και στη γραφική παράσταση ότι 30.000 με 45.000 νέες θέσεις εργασίας δημιουργούνται χάρη στην επένδυση στις ε, νέες υπηρεσίες περίθαψης παιδιών. Έγινε πρόσφατα μελέτη λοιπόν όπως σας είπα στην Αυστρία θα ήταν ενδιαφέρον να γίνει μια ολιστική μελέτη κόστους ωφέλους και σε άλλες χώρες όσον αφορά το πόσο επιδρά η δημιουργία νέων κέντρων περίθαλψης παιδιών. Βλέπετε ότι η φροντίδα των παιδιών και άλλων εξαρτημένων συγγενών είναι ένας στους βασικούς λόγους για εκείνους που δεν μπορούν να απασχοληθούν ή να δουλέψουν όσο θα θέλαν. τόσες ώρες όσο θα θέλαν. Τονίσαμε τους στόχους της Βαρκελόνης όσον αφορά τη διαθεσιμότητα κέντρων φροντίδας παιδιών και ίσως λόγω μέτρων λιτότητα σε κάποιο βαθμό και λόγω της κρίσης είχαμε διάφορα διάφο, αντίκτυπο όσον αφορά τα τέλη που ζητούνται σύμφωνα με τις μελέτες το κόστος είναι ο μεγαλύτερος φραγμός για την πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες φροντίδας παιδιών. Και αν το προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε ή να βοηθήσουμε τους νέους να μπουν στην αγορά εργασίας, είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη όχι μόνο το κόστος των υπηρεσιών φροντίδας παιδιών, αλλά να δούμε και ποιες είναι οι συνέπειες των μεταρρυθμίσεων, ε, των διάφορων φορολογικών μεταρρυθμίσεων όσον αφορά το επίπεδο διαβίωσης των μελών της οικογένειας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω πως πραγματικά καταστήσατε σαφή τη σημασία της ε, παιδικής μέρημνας. Πιστεύω πως η φροντίδα των παιδιών είναι ένα από τα σημεία κλειδιά εδώ. Έχει να κάνει και με την οικονομική ανεξαρτησία έτσι κι Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση μάλιστα σε σχέση με την υποδομή. Τώρα θα σας δώσω την δυνατότητα να λάβετε το λόγο. Κυρία Μορβάη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Σημείωσα ότι χρησιμοποιούσατε μια ουδέτερη ως προς το ε, φιλογλώσσα όταν κάνατε λόγο για τις επιπτώσεις της παιδικής εμέριμνας και του συστήματος παιδικής εμέριμνας στην απασχολησιμότητα των ανθρώπων, όπως είπατε. Είναι πολύ αισιόδοξο το σενάριο που παρουσιάσατε και πιστεύω ότι ειδικά τώρα δεν ισχύει αυτό, ότι αφορά και πλήττει τις γυναίκες πολύ περισσότερο από ό,τι τους άνδρες. Και παρακαλώ διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά πιστεύω ότι οι γονεϊκές ευθύνε είναι πρωτίστως ε, κάτι ιδίων των γυναικών, όπως θεωρείται σε πολλά μέρη της Ευρώπης. Όπως για παράδειγμα στη δική μου χώρα, που έχει κομμουνιστικό παρελθόν, ή ενδεχομένως και σε κάποιες χώρες στη Νότια Ευρώπη. Οι γυναίκες επομίζονται το βάρος της ε, ανατροφής των παιδιών μόνες τους. Και αυτό σαφώς και επηρεάζει τις ευκαιρίες που έχουν, τις δυσκολίες όπως ε, ακούσαμε και πιο πριν, πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Η πρώτη ερώτηση που κάνουν οι εργοδότες είναι έχετε παιδιά, σκοπεύετε να κάνετε, πότε σκοπεύετε να κάνετε. Και αυτό προφανώς δυσχεραίνει την κατάσταση για τις γυναίκες. Το ερώτημα λοιπόν που έχω να θέσω είναι, θα αλλάξει καθόλου αυτό θα αλλάξει η απασχολησιμότητα και των ανδρών, εάν λάβουμε υπόψη αυτόν τον παράγοντα. Και αυτός ο παράγοντας, η γονεϊκή ευθύνη αφορά τους άνδρες. Θα αλλάξει κάτι στις εγκαταστάσεις φροντίδας ε, παιδιών Αυτέ οι εγκαταστάσει, παιδική σταθμή α πούμε, θεωρούνται κοινό αγαθό, δημόσιο αγαθό ή θεωρούνται κάτι που θεωρείται κάτι πρέπει να αναλάβουν αποκλειστικά οι γυναίκες. Εάν η φροντίδα αποκλειστικα οι γυναικες εαν η φροντιδα ανατροφη των παιδιών είναι κοινή ευθύνη ανδρών και γυναικών, πώς αυτό θα αλλάξει την ισορροπία δουλειά και οικογένεια στον εργασιακό χώρο. Δηλαδή, θα υπάρξει κάποια σαφή ε, ρύθμιση, θα γίνει κατανοητό ότι κάποιε ώρε θα είναι αφιερωμένε αποκλειστικά και μόνο στη δουλειά, κάποιες άλλε, αποκλειστικά και μόνο στην οικογένεια και στην ευθύνη ανατροφή. Πώ αυτό συνδέεται με το όλο ζήτημα της, ε, των εγκαταστάσεων, ε, των παιδικών σταθμών, α πούμε, παιδική μέρημνα. Πιστεύω πω είναι ένα στοιχείο πολύ σημαντικό για να επιτευχθεί ισότητα ανδρών και γυναικών. Περίπλοκα τα έθεσα, αλλά αυτό ήθελα να ρωτήσω. Παρακαλώ. Όπως Ας το δούμε λοιπόν μέρος μέρος. Καταρχάς όσον αφορά την... τον επιμερισμό των καθηκόντων στο σπίτι. Βλέπουμε τα στοιχεία της ε, μελέτης. Βλέπουμε λοιπόν από αυτά ότι οι γυναίκες συνεχίζουν να περνάνε περισσότερη ώρα φροντίζοντας τα παιδιά τους στο σπίτι. Επίσης ε, σε μια μελέτη για τις συνθήκες εργασίας ε, βλέπουμε μια αλλαγή στις τάσεις τα πιο πρόσφατα δεδομένα που έχουμε μας δείχνουν ότι τώρα έχει τροποποιηθεί λίγο το μοντέλο του κουβαλητή στο, σε ένα σπιτικό, σε ένα νοικοκυριό. Υπάρχει ένας που έχει μία δουλειά πλήρους απασχόλησης και ο δεύτερος ενήλικας έχει μία δουλειά μια απασχόλησης. Κάποιες άλλες αλλαγές που έχουμε παρατηρήσει στην άτυπη φροντίδα, στη φροντίδα στο σπίτι δηλαδή, στην ανατροφή των παιδιών, είναι ότι συμμετέχουν και οι παππούδες και οι γιαγιάδες, όλο ένα και περισσότερο. Ο του τους ε, γίνεται όλο ένα και σημαντικότερος ε, στην παροχή επίσημης φροντίδας σε ένα νοικοκυριό. Μάλιστα δημοσιεύτηκε μία μελέτη με τίτλο «Οι παππούδες και οι γιαγιάδες σώζουν το νοικοκυριό σε χώρες, για παράδειγμα, όπου η παιδική μέρημνα δεν είναι τόσο ανεπτυγμένη όπως σε χώρες της Νότιας Ευρώπης. Οι γιαγιάδες λοιπόν και οι παππούδες φροντίζουν τα παιδιά, ενώ οι γυναίκες εργάζονται. Τώρα, όσον αφορά το ρόλο των ε, υπηρεσιών παιδικής μέρημνας και το πώς αυτές σχετίζονται με τα ζητήματα της ισότητας των φίλων. Πιστεύω πως αυτές οι εκτιμήσεις που έχουμε από το επιμελητήριο εργασίας μας δείχνουν μεν κάποια στοιχεία, κάποια νούμερα, αλλά μας δείχνουν και τις επιπτώσεις στην οικονομία σε γενικές γραμμές. Δηλαδή τις ετάσεις της ε, στον ε, κλάδα των κατασκευών, για παράδειγμα, όπου κυριαρχούν οι άνδρες, μας δείχνουν τις ε, αυξητικές τάσεις στην, στους ε, τομείς αυτούς, στην φροντίδα των παιδιών και φυσικά η συμπερίληψη των γυναικών στην αγορά εργασίας σε αυτούς τομείς είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό Και η δημιουργία αυτών των λεγόμενων νέων θέσεων εργασίας 30 45.000 είναι κάτι που θα επιταχύνει την συμπερίληψη των γυναικών. Θα, θα αυξηθούν μεν οι ώρες εργασίας, θα αυξηθεί βέβαια και η κατανάλωση. Μάλιστα. Ευχαριστώ για μία ακόμα φορά. Κύριε μονινούέβο, για τη συμμετοχή σας στο συνέδριο αυτό. Θα προχωρήσουμε τώρα στον επόμενο ομιλητή στην επόμενη παρέμβαση και ο τελευταίος αυτού του πάνελ, ο Ματίας Σούτερ από το Πανεπιστήμιο του Ίνσπρουκ και το Πανεπιστήμιο του Γκέτεμπορ. Θα μας παρουσιάσει λοιπόν τα αποτελέσματα της έρευνάς του σχετικά με τις διαφορές ανδρών και γυναικών στην προθυμία ανταγωνισμού, στα, στις αιτίες και στα αποτελέσματα των παρεμβάσεων. Ματίας είναι καθηγητής πειραματικής οικονομίας και μελετά το πώς ε, αναπτύσσεται η οικονομική συμπεριφορά. Ευχαριστώ πολύ. Όταν μιλάμε για διαφορές ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας, καταρχάς το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μεγαλύτερο ενδιαφέρον από πλευράς των ανδρών. Και αυτό έχει σχέση με αυτό που θα σα πω. Εάν δεν έχετε αντιληφθεί μέχρι τώρα ότι υπάρχουν διαφορές στην αγορά εργασία σε άντρε και γυναίκες, μισθολογικέ, διαφορές στην προαγωγή, τότε μέχρι το τέλος αυτού του συνεδρίου θα έπρεπε να το έχετε συνειδητοποιήσει. Υπάρχουν κάποιες επεξηγήσεις. Ορισμένες τις έχουμε αναφέρει σήμερα, για παράδειγμα, τι διακρίσει. Απλή και ξεκάθαρη διάκριση εις βάρος των γυναικών. Επίσης, μια άλλη παραδοσιακή επεξήγηση είναι τα προβλήματα που δημιουργούν ένα περιβάλλον στο οποίο οι γυναίκες δεν μπορούν εύκολα να συνδυάσουν καριέρα και οικογένεια. Ε, ορισμένοι κλάδοι της οικονομίας είναι εχθρικοί για τις γυναίκες, για παράδειγμα. Ορισμένοι τομείς ε, στους οποίους η συμμετοχή των γυναικών μειώνεται σταδιακά. Σε αυτό που θέλω να επικεντρωθώ εγώ είναι κάτι που έχουμε παρατηρήσει σε στην πανεπιστημιακή κοινότητα τα τελευταία 10-15 χρόνια. Είναι κάτι, ένας επιπρόσθετος παράγοντας στις διαφορές ανδρών και γυναικών. Ποιος είναι αυτός λοιπόν διαφορά στην προθυμία ανταγωνισμού και στην προθυμία του να εκτεθείς στον ανταγωνισμό. Αυτό σίγουρα είναι πολύ σημαντικό. Και ας δούμε τώρα τι γίνεται. Ας προσπαθήσουμε. Είναι κάτι ίσως που δεν πρέπει να διαβάσετε να βλέπετε τις, διαβα... τις διαφάνειες. Πείτε μου, σηκώστε το χέρι εάν πήρατε τη δουλειά σας χωρίς να ανταγωνιστείτε κανέναν. Πείτε μου λοιπόν αν πήρατε τη δουλειά σας χωρίς ανταγωνισμό. Α, εσείς το κάνατε. Τέλεια. Είστε εξαίρεση όμως. Είναι κάτι που χρησιμοποίησα για να σας δείξω ότι αν δεν γνωρίζουμε μια κατάσταση αν δεν, είμαστε, αν δεν αισθανόμαστε άνετοι σε ένα περιβάλλον ανταγωνιστικό, δεν έχουμε να κερδίσουμε τίποτα. Τώρα, Εάν δεχτούμε ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες όσον αφορά την προθυμία ανταγωνισμού, αυτό θα έχει πολύ μεγάλες συνέπειες στα επιχειρήματά μας. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία μας δείχνουν ότι οι γυναίκες δύσκολα θα μπουν σε ανταγωνισμό, πιο δύσκολα από ότι οι άνδρες. Και αυτό τους επηρεάζει στους μισθούς, τους επηρεάζει στις προαγωγές αργότερα. Και υπάρχουν αποδείξεις ότι αυτό ισχύει και για τους ενήλικες. Και αυτό μας δημιουργεί δύο ερωτήματα. Το πρώτο είναι τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Και αυτό μας οδηγεί αμέσως στην επόμενη ερώτηση. Ερώτηση, δηλαδή, οποιαδήποτε μορφή παρέμβαση, ποια στοιχεία θα έχει. Και εδώ θα έρθω στο δεύτερο μέρος της παρουσίασής μου. Να σας πω όμως ότι μία παρέμβαση πολιτικής δεν πρέπει να αρχίσει χωρίς να έχει λάβει ε, ε, επίγνωση αυτών των διαφορών και των που προκαλούν. Διότι, εάν θέλουμε να κάνουμε μια σωστή πολιτική, πρέπει φυσικά να έχουμε απόλυτη επίγνωση τη κατάσταση στην όπου παρατηρούνται συμπεριφορικές διαφορές ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες. Γιατί αυτές θα μας δείξουν και το χρονικό σημείο το οποίο είναι πιο κατάλληλο να παρέμβουμε. Και αυτό θα είναι το πρώτο μέρος της ομιλίας μου σήμερα. Και μια από πολλές οι παρουσιάσεις έτσι μας έδωσαν αυτά τα νούμερα, τα, τις, τα χώρισαν σε ηλικιακές ομάδες, ήταν πολύ λεπτομερείς. Εγώ θα συνεχίσω έτσι, αλλά θα κατέβω ηλικιακά, θα πάω στα τρίχρονα, σε ηλικία παιδικού σταθμού. Και θα δείτε τι θέλω να πω. Ας μπούμε λοιπόν στο ψητό. Θα σας παρουσιάσω λοιπόν κάτι το οποίο είναι μία έρευνα σε πολύ προσωπικό επίπεδο. Είναι μία πειραματική μελέτη, ένα πείραμα, το οποίο συμπερίλαβε περίπου πάνω από 1.500 παιδιά από 3 έως 18 ε, χρονών. Τους ε, έβαλαν να κάνουν τρία πράγματα. Ε, να τρέξουν, να κάνουν μαθηματικές πράξεις και να πάρουν πράγματα από ένα καλάθι. Και εκεί παρατηρήσαμε πάρα πολλές διαφορές όσον αφορά την προθυμία να ανταγωνιστούν. Ας αρχίσουμε λοιπόν. Θα το κάνω με χρονολογική σειρά για να δείτε τι εννοώ. Το πρώτο λοιπόν που κάναμε, πήραμε εφήβους. Μια και έχουμε αποδείξει σε ενήλικες ότι οι γυναίκες ε, δεν προτιμούν τον ανταγωνισμό, σκεφτήκαμε και είπαμε ας δούμε τι γίνεται και με τους εφήβους, αν ισχύει αυτό και για αυτού. Γι' αυτό λοιπόν πήγαμε σε παιδιά 9 έω 18 χρονών και είχαν κάποιους διψήφιους αριθμούς. Έπρεπε να τους επιλέξουν, ήταν τελείω τυχαίοι και μετά πληρώθηκαν. Αυτό λοιπόν ήταν η προϋπόθεση. Τους πληρώνονταν ανάλογα με τη δουλειά που έκαναν. Και να σας πω ότι τα άτομα αυτά δεν ήταν τελείως αδιάφορα ως προς το χρήμα. Δεν το θεωρούσαν παιχνίδια. Έχουμε αποδείξεις ότι τους ενδιέφερε λοιπόν η αμοιβή. Αυτό που έπρεπε να κάνουν ήταν πάρα πολύ απλό. Έπρεπε να προσθέσουν λοιπόν αυτά τα διψήφια νούμερα και αν είσαι γρήγορος μπορείς να βρεις πολύ γρήγορα το αποτέλεσμα και μετά μπορούσες να επιλέξεις εάν θέλεις να πληρωθείς με βάση τις σωστές σου απαντήσεις ή με βάση εναλλακτικά με βάση τη θέση που έχεις απέναντι στους συναγωνιστές σου, στους ανταγωνιστές σου μάλλον, συγγνώμη. Δηλαδή, αν είσαι ο καλύτερος, θα πάρεις περισσότερα. Αν χάσεις δεν θα πάρεις τίποτα. Έτσι λοιπόν είχαν την επιλογή είτε να πάρουν τέσσερις φορές περισσότερα χρήματα από τους υπόλοιπους είτε να πληρωθούν ανάλογα με το τι κάνουν. Δηλαδή αυτό στις κανονικές συνθήκες εργασίας τι, τι, ε, με, με τι αναλογεί. Αναλογεί με μια πολύ ανταγωνιστική θέση εργασίας. Και αυτό που είδαμε τι ήταν ότι εδώ βλέπετε τις πέντε διαφορετικές ηλικιακέ ομάδες. 9, 10, 11, 12, 13, 14 και ούτε καθεξής. Οι σκοτεινέ μπάρε είναι πάντα οι άνδρες και δείχνουν τι σωστέ απαντήσει και η ανοιχτόχρωμη μπάρα είναι πάντα γυναίκε. Έχουμε λοιπόν αυτό. Πρώτον, βλέπουμε είναι ε, ότι σταδιακά με την ηλικία ε, γίνονται καλύτεροι και μπορούν να απαντήσουν καλύτερα. Άρα λοιπόν κάτι μαθαίνουν στο σχολείο, βλέπουμε. Και αυτό λοιπόν είναι, μια, είναι κάτι που μπορούμε να, να χρησιμοποιήσουμε για να προβλέψουμε τη μελλοντική τους, τις μελλοντικές τους απολαβές. Έπειτα, οι αγγίλες μας δείχνουν το εξή. Μας δείχνουν ότι η διαφορά ανδρών και γυναικών δεν είναι, είναι αμεληταία, ότι είναι εξίσου καλή σε αυτό που κάνουν. Αυτό βλέπουμε ότι ισχύει για όλες τις ηλικιακές ομάδες. Τώρα, όσον αφορά την απόδοση και την επιθυμία και την θέληση ανταγωνισμού, στην στο επόμενο γράφημα βλέπετε πόσο πιθανό είναι να διαλέξουν οι άνδρες ή οι γυναίκες το... την πληρωμή την ανταγωνιστική. Και εδώ θα δείτε ότι η μπάρα που δείχνει τους άνδρες είναι διπλάσια από την μπάρα των γυναικών. Δηλαδή, οι γυναίκες, τι σημαίνει αυτό, δεν θέλουν να ανταγωνίζονται. Επιλέγουν να μην μπουν σε αυτή την θέση. Είναι πραγματικά εκπληκτικά τα αποτελέσματα και είναι ανησυχητικά θα έλεγα, διότι βλέπουμε ότι τα προσόντα δεν παίζουν ρόλο εδώ πέρα, αλλά παίζουν ρόλο τα στερεότυπα. Αλλά θα επιστρέψω σε αυτό. Θέλετε να διακόψετε, παρακαλώ. Μάλιστα. Δεν επιτρέπεται να διακόψει η συνάδελφος. Καλά, θα δεχτώ ερωτήσεις σε κάθε περίπτωση. Τώρα, ίσως πιστεύετε ότι αυτά που κάνουμε εδώ δεν θα έχουν σημασία σε βάθος χρόνου. Έτσι λοιπόν, για να, το κοιτάξουμε, για να κοιτάξουμε και εμείς αυτό, γιατί και εμείς θέλαμε να το κοιτάξουμε, επανήλθαμε. Τους ερωτήσαμε μετά από δύο χρόνια, κάναμε το ίδιο πείραμα και είχαμε ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα. Θέλαμε δηλαδή να δούμε εάν θα είσαι ανταγωνιστικό σήμερα και δεν θα είσαι ανταγωνιστικό σε δύο χρόνια. Δεν ίσχυε. Οι τάσει βέβαια που παρατηρήσαμε ήταν ότι οι γυναίκε που συμμετείχαν στον ανταγωνισμό μετά από δύο χρόνια δεν είχαν ε, τόσο έντονη επιθυμία, ενώ οι άντρε αντίθετα είχαν αυξημένη επιθυμία. Αυτό που κάναμε τώρα με τους εφή... αυτό το ήταν που κάναμε με τους εφήβους. Τώρα πήγαμε πιο κάτω, πήγαμε σε παιδιά. Είχαμε δύο πράγματα που έπρεπε να κάνουν. Έπρεπε να τρέξουν 30 μέτρα στο γυμναστήριο και αυτό που είχαν να επιλέξουν ήταν είτε θα το κάνεις μόνος σου είτε θα τρέξεις με κάποιον άλλο που έχει επιλεγεί τυχαία. Ανταγωνισμός δηλαδή. Ποιος θα έρθει πρώτος, ποιος θα νικήσει. και πάλι είχαμε διαφορετικά κίνητρα. Δηλαδή, αν επέλεγε τον ανταγωνισμό, φυσικά μπορούσε να κερδίσει τα διπλάσια από ό,τι έτρεχε μόνο σου, αλλά αν έχανε, δεν έπαιρνε τίποτα. Και αυτό, μάλιστα, σε αυτέ τις ηλικίε είναι και αιτία για να βάλει κανεί τα κλάματα. Τι είδαμε λοιπόν. Βλέπουμε την απόδοση βλέπουμε τον χρόνο που χρειάστηκαν για να τρέξουν αυτή την απόσταση, τα, ε, και οι ομάδε 3, 4, 5, 6 και 7, 8. Και φυσικά, ναι, ωραία, το προφανές είναι ότι όσο μεγαλώνεις γίνεσαι και ταχύτερος. Και δεν, υπάρχει, ε, δεν υπάρχουν εδώ διαφορές στην ε, ταχύτητα ανδρών και γυναικών. Και να σας πω ότι οι σωματικές διαφορές ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες αρχίζουν στην εφηβεία σε αυτές τις ηλικίε στο 5 έως 6 χρονών, δεν υπάρχουν σωματικές διαφορές ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες, στις επιδόσεις, στην ταχύτητα. Μετά στο δεύτερο γράφημα βλέπουμε την προθυμία να ανταγωνιστούν. Και εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι παρότι είναι το ίδιο γρήγοροι άνδρες και γυναίκες, αγόρια και κορίτσια, τα αγόρια επέλεξαν περισσότερο από τα κορίτσια να ανταγωνιστούν, να τρέξουν μαζί με κάποιον άλλον. Όπω σα ε, είπα και σα ε, επαναλαμβάνω, δεν έχει να κάνει με τι ικανότητε αυτό. Υπάρχουν μελέτε επιστημονικέ που έχουν δείξει ότι οι αγόρια και οι κορίτσια σε αυτές τι ηλικίε έχουν ακριβώ τι ίδιε δυνατότητε. Τώρα, κάτι άλλο που έπρεπε να κάνουν, το οποίο ήταν πιο ευνοϊκό για τα κορίτσια. Αριστερά βλέπετε ένα καλάθι με πολλά διαφορετικά αντικείμενα. Αυτό που έπρεπε να κάνουν λοιπόν είναι από το γαλάζιο καλάθι να μαζέψουν όλα τα κυλινδρικά αντικείμενα και να τα βάλουν στο ποτήρι Ξέρουμε από την ψυχολογία ότι οι γυναίκες είναι καλύτερες από την εξελικτική ψυχολογία ότι οι γυναίκες είναι καλύτερες σε αυτές τις εργασίες από μικρότερη ηλικία. Αυτό δηλαδή λοιπόν το τεστ ήταν περισσότερο ευνοϊκό για τις γυναίκες, για τα κορίτσια. Θέλαμε λοιπόν να δούμε εάν ισχύει αυτό, εάν τα κορίτσια θα έχουν καλύτερα αποτελέσματα και αν αυτό θα επηρεάσει την προθυμία να ανταγωνίζονται, να ανταγωνιστούν. Γι' αυτό λοιπόν τι κάναμε. Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον όπου όλα τα κορίτσια είχαν ευνοϊκότερες συνθήκες αντιμετώπισης από ότι τα αγόρια. Δηλαδή και ήταν καλύτερες αυτό που έπρεπε να κάνουν και είχαν ευνοϊκότερε συνθήκες και θέλαμε να δούμε εάν θα συνέχιζαν να έχουν την ίδια επιθυμία ανταγωνισμού ή αν αυτή θα είχε αυξητικέ σημειωτικές τάσεις. Αυτό, δηλαδή τους δώσαμε ένα προβάδισμα 2 προς 1. Εδώ βλέπουμε τον, ε, τον ανταγωνισμό, τα ποσοστά για τα τρίχρονα και τα τετάχρονα δεν βλέπουμε διαφορές ε, σε αγόρια και κορίτσια και αυτό είναι καλό. Δηλαδή αυτά τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίε δεν παρουσιάζουν διαφορές στην προθυμία ανταγωνισμού. Όμως από την ηλικία των 5-6 χρόνων και μετά το παιχνίδι έχει τελειώσει. Βλέπουμε ότι ακόμα και σε, ένα, ε, και σε κάτι στο οποίο τα κορίτσια είναι καλύτερα από ότι τα αγόρια, τα κορίτσια αποφεύγουν τον ανταγωνισμό και τα αγόρια τον προτιμούν πολύ περισσότερο. Ποιε είναι λοιπόν οι αιτίε πίσω από αυτό. Καταρχάς υπάρχει βέβαια διαφορά, υπάρχει χάσμα ανάμεσα στα δύο φύλλα. Γιατί βλέπουμε καταρχάς και μπορούμε να το μετρήσουμε ότι οι γυναίκες αποφεύγουν περισσότερο τον κίνδυνο και ο ανταγωνισμό φυσικά και συμπεριλαμβάνει κινδύνους. Υπάρχουν και βιολογικές εξηγήσει για το ότι γιατί οι γυναίκες αποφεύγουν τον ανταγωνισμό. Το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι τα αγόρια έχουν υπερβολική αυτοπεποίθηση περισσότερο από ό,τι τα κορίτσια. Όταν τους ρωτήσαμε για τις επιδόσεις τους, οι γυναίκες είχαν μια σχετικά καλή επίγνωση του πώς τα πήγαν, ενώ τα αγόρια είχαν ε, θεώρησαν πως τα πήγαν καλύτερα από ό,τι τα πήγαν. Μπορεί να γελάτε, αλλά αυτό ήταν. Ήταν αλήθεια, αλήθεια αυτό. Και αυτό πραγματικά συνεισφέρει στην διαφορά, στο χάσμα ανδρών και γυναικών. Και βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει κάτι και δεν ξέρουμε τι είναι. Μπορεί να είναι λοιπόν στερεότυπο, μπορεί να είναι η εκπαίδευση, η παιδεία, δεν το ξέρουμε. Είναι όμως, η... είναι όμως προφανές. Έχουμε τις αποδείξεις. Τώρα, αυτό ολοκληρώνει το πρώτο μέρος του τεστ και ήταν πάρα πολύ σημαντικό γιατί τι μας έδειξε ότι αν δούμε, αν το μεταφέρουμε αυτό στην αγορά εργασίας θα δούμε ότι ένας τουλάχιστον παράγοντας που συμβάλλει στις διαφορές ανδρών και γυναικών ε, αρχίζει πολύ πιο νωρίς από ότι η ηλικία εισόδου στην αγορά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για οποιαδήποτε πολιτική θέλουμε να χαράξουμε, για οποιαδήποτε σχέδιο θέλουμε να καταστρώσουμε. Τώρα, πώς μπορούν να ε, είναι καρποφόρες οι παρεμβάσεις της πολιτικής. Εδώ κάναμε ένα άλλο πείραμα με φοιτητές, με πανεπιστημιακούς φοιτητές, όπου φυσικά θέλαμε και πάλι να μετρήσουμε το πόσο θέλουν να συμμετέχουν σε ανταγωνισμό. Είχαμε 360 φοιτητές και τους χωρίσαμε σε ομάδες 6 ατόμων, τρεις άνδρες, τρεις γυναίκες σε κάθε ομάδα και η κάθε ομάδα θα έχει δύο νικητές. Δηλαδή ο ανταγωνισμός είναι ανάμεσα σε μία ομάδα τρει άνδρες, τρει γυναίκες με δύο νικητέ σε κάθε ομάδα. Εδώ δεν είχαμε την ίδια αντιμετώπιση από ό,τι με τα μικρότερα παιδιά. Είχαμε πέντε προϋποθέσεις ε, τις οποίες χρησιμοποιήσαμε. Καταρχάς ο έλεγχος. Οι δύο νικητές είναι τα μέλη της ομάδας που είχαν τις καλύτερες επιδόσεις. Και αυτό είναι πολύ εύκολο να το μετρήσουμε. Δεύτερο, η αυστριακή μεταχείριση, όπως θέλω να την αποκαλώ, η επανάληψη του τουρνουά. Δηλαδή, εάν και οι δύο νικητές είναι άνδρες, τότε επαναλαμβάνεται ο διαγωνισμός. Και μπορούμε δηλαδή να κάνουμε reboot και να αρχίσουμε από την αρχή. Αυτό έχει και πολιτικό σκεπτικό. Αυτοί λοιπόν οι δύο παράγοντες ήταν οι πιο σημαντικοί. Τρία, ελάχιστες ποσοστώσεις, δηλαδή τουλάχιστον μία γυναίκα στους δύο νικητές. Και η γυναίκα με τις καλύτερες επιδόσεις πάντα κερδίζει. Τρίτη λοιπόν επιλογή. Τέταρτη επιλογή, προτιμησιακή μεταχείριση τα γνωρίζετε όλα αυτά. Δηλαδή, αν κάποιοι έχουν ίσα προσόντα, οι γυναίκες θα έχουν προτιμησιακή μεταχείριση. Έτσι λοιπόν, το εφαρμόσαμε αυτό και δώσαμε έναν πόντο προβάδισμα σε κάθε γυναίκα της ομάδας. Αυτό δηλαδή που λέμε προτιμησιακή μεταχείριση. Μπορούμε να το κάνουμε και ακόμα πιο έντονο, το παρακάνουμε ενδεχομένω. Η προτιμησιακή συμπεριφορά 2. Του δίνουμε τόσο μεγάλο προβάδισμα, ώστε ακόμα και γυναίκε με πολύ χαμηλέ επιδόσει μπορούν να ξεπεράσουν του άντρε. Εδώ δηλαδή το παρατραβήξαμε λιγάκι. Τι είδαμε. Κοιτάξτε αυτή τη διαφάνεια, αυτή την πλευρά. Εδώ πέρα είναι ο έλεγχος, το πλασέμπο δηλαδή. Εδώ πέρα βλέπετε την ανδρική συχνότητα επιλογής ανταγωνισμού, πολύ μεγαλύτερη από ότι των γυναικών. Αυτά τα ξέρετε ήδη, σας τα, τα έχετε ακούσει. Τώρα, ας πάμε στην δεξιά πλευρά. Η αυστριακή συμπεριφορά, η αυστριακή μεταχείριση, σαρκαστικά το λέω, δεν έχει καμία απολύτως, καμία απολύτως ε, Κάνει απολύτω αποτέλεσμα. Α δούμε τώρα τι γίνεται στη μέση. Εάν έχουμε ελάχιστε ποσοστώσει με, προ... με πρημοδότηση των γυναικών σε περίπτωση ισοπαλία, θα δούμε ότι δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε άντρε και γυναίκε όσον αφορά την προθυμία έκθεση σε ανταγωνισμό. Και αυτό ακριβώ θέλουμε να κάνουμε με τις πολιτικές μας παρεμβάσεις. Και αυτό που δεν μπορείτε να δείτε πίσω από τα γραφήματα είναι ότι οι γυναίκες που ενθαρρύνονται να συμμετέχουν στον ανταγωνισμό είναι αυτές με τις καλύτερες επιδόσεις. Δεν θέλουμε δηλαδή να πρημοδοτήσουμε γυναίκες με χαμηλά προσόντα. Όχι, αυτό ας το ξεκαθαρίσουμε. Αυτές οι παρεμβάσεις θέλουν να δώσουν κίνητρα στις γυναίκες με τις καλύτερες επιδόσεις να εισέλθουν στον ανταγωνισμό και να μην τον αποφεύγουν. Και αυτό είναι κάτι με πολύ μεγάλη σημασία, διότι πραγματικά δεν θα έπρεπε να μας ενδιαφέρει το φίλο, αλλά ποιος είναι ο καλύτερος. Έχω άλλα δύο λεπτά, οπότε θα ολοκληρώσω μέσα σε αυτά. Ανταγωνισμό λοιπόν υποπίεση. Ο ανταγωνισμό υποπίεση είναι κάτι που οι γυναίκε δεν επιθυμούν, δεν του αρέσει, αρχίζει από τον υπηαγωγείο, αρχίζει από την υπηακή λοιπόν ηλικία ακόμα και σε πράγματα στα οποία οι γυναίκε είναι καλύτερε. Αυτή τη στιγμή σκοπεύουμε να αρχίσουμε ένα project σύμφωνα με το οποίο θα μελετήσουμε βιολογικές επιτυχίες του ανταγωνισμού Υπάρχουν και άλλες έρευνες που πρέπει να κάνουμε. Αυτό λοιπόν δρομολόγουν έπειτα. Το χάσμα ανάμεσα στα φύλλα συνεχίζεται μέχρι τα 18 χρόνια και επιμένει και ανάμεσα στους ε, ανθρώπους. Δεν μπορείς λοιπόν δηλαδή να στοχεύσεις σε μια ιδιαίτερη πληθυσμιακή ομάδα, σε γυναίκες δηλαδή με πολύ υψηλά προσόντα. Και τέλος, ή θετική δράση. Οι πολιτικές δηλαδή με τι ελάχιστε ποσοστώσει με την προτιμησιακή μεταχείριση μπορούν να βοηθήσουν ως, ε, προς το να οθήσουν τις γυναίκες στον ανταγωνισμό, τις γυναίκες με τις καλές επιδόσεις και έχουμε αποτελέσματα. Ιδιαίτερα αν τα μεταφέρω αυτά σε μια πολιτική μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα. Και το ερώτημα που δημιουργείται τώρα είναι αν αυτές οι θετικέ δράσεις θα έχουν αποτελέσματα. Να σας πω ότι καταρχάς πρέπει να γίνουν διεξοδικές έρευνες προτού εφαρμοστεί κάτι τέτοιο. Και να σας πω ότι δεν είναι όλες από αυτέ τέλειες. Εμείς βέβαια στην Αυστρία έχουμε τέτοιε πολιτικέ, έχουμε καλά αποτελέσματα, αλλά δεν μπορώ να πάρω όλο όλα τα εύσημα. Δεν είμαστε η μόνη χώρα με καλά αποτελέσματα. Αυτά λοιπόν. Ελπίζω να μην σα κούρασα και να απολαύσετε και τις επόμενες παρεμβάσεις. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι να αρχίζουμε καιρός, να μην καθυστερούμε ε, Επίση, είναι πολύ δύσκολο να πιστεύουμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε τα πάντα όσα ισχύουν σε σχέση με τα στερεότυπα σε πανεπιστημιακό επίπεδο ή και νωρίτερα. Σα ευχαριστούμε. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα στοιχεία. Ε, κυρία Μορβάη, θα κάνει την πρώτη ερώτηση. Ευχαριστώ. Τα ευρήματα τη έρευνα σα, όντω θα πρέπει να αληθεύουν διότι μόνο ακούγοντας ε, όλα αυτά που είπατε για τον ανταγωνισμό κουράστηκα. Ε, μάλλον επειδή είμαι γυναίκα. Εξαντλήθηκα. Πάντως, ε, αν απορρίπτουν οι γυναίκες αυτόν τον διαρκή ανταγωνισμό στη ζωή και επιλέγουν την οδό της συνεργασίας αντί του ανταγωνισμού για να νιώθουν γυναίκες, αναρωτιέμαι. Όχι ότι αυτό είναι απαραίτητα ο στόχος της ομιλίας σας, αλλά εγώ αναρωτιέμαι για ποιο λόγο Οι παραδοσιακά αντρικές αξίες στη ζωή, όπως ο ανταγωνισμός, θεωρούνται ανώτερες και εμείς θα πρέπει και να το δεχτούμε και να μάθουμε να γίνουμε πιο ανταγωνιστικές κατά τη διαστολή με την άλλη εναλλακτική λύση να μάθουν να συνεργάζονται περισσότερο οι άντρες παραδείγματο χάρη να μην χρειάζονται ένα διαρκή ανταγωνισμό στον πολιτικό βίο είναι ξεκάθαρο αυτό πόσο επιζήμιο είναι να θεωρείται ως ύψιστη αξία ε, αυτό το πνεύμα ανταγωνισμού αντίστα με την συνεργασία. Αυτά γίνονται στην πολιτική, ανταγωνίζονται τα κόμματα, μεταξύ τους αρνούνται να συνεργαστούν ώστε να αντιμετωπίσουν ένα οποιοδήποτε ζήτημα κοινωνικό ή άλλο και να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να επιλύσουν ε, ένα τέτοιο πρόβλημα. Δεν θα ήταν πιο λογικό και στην οικονομία τα ίδια γίνονται επικρατεί ο ανταγωνισμός ε, και η καταπίεση των αδυνάτων ε, αντί να επικρατήσει η συνεργασία και να επικρατήσει η κοινωνική ε, δικαιοσύνη, να νιώθουν όλοι ότι έχουν ένα στόχο και έχει ένα νόημα η ζωή τους. Ε, με τα συμπεράσματα που αντλήσατε εσείς θα συμφωνήσω όμως ε, όλο αυτό το ζήτημα του ανταγωνισμού και ότι απαραίτητα πρέπει να θεωρείται ως ύψιστη αξία σε σχέση με την αντίθετη έννοια της συνεργασία. Εγώ δεν νομίζω ότι αληθεύει αυτό. και οι αντρικές αξίες ε, δεν είναι θέσφατες και ίσως αν μετατοπιστούμε από τις παραδοσιακές αντρικές αξίες προς τις ε, παραδοσιακά γυναικείες αξίες, ίσως να φτιάξουμε και ένα καλύτερο κόσμο. Απάντηση. Το αντιλήφθην ε, το νόημα της παρέμβασής σας, σας διαβεβαιώ ότι το μεγαλύτερο τμήμα της έρευνάς μας επικεντρώνεται γύρω από την έννοια της συνεργασίας. Να με καλέσετε στο επόμενο εργαστήρι για τις ε, διαφορές στα δύο φύλλα ως προς την ε, συνεργατική συμπεριφορά σε ομάδες, γιατί είναι και ένας από τους τομείς που ερευνώ προσωπικά. Πρώτα απ' όλα ε, θα ήταν πλήρης παρανόηση αν επιστρέψετε και σκεφτείτε ότι ο Ματίας ε, Στάρκε ισχυρίστηκε ότι είναι ανώτερα τα ανδρικά ιδανικά. Ε, δεν θα ήθελα να αποχωρήσετε με αυτή την εντύπωση γιατί δεν αληθεύει. Ποιο όμως είναι το θέμα πώς βλέπω εγώ τον κόσμο και πώς τον βλέπουν οι άλλοι. Για πολλές θέσεις έχει ιδιαίτερη σημασία να είναι κανείς ανταγωνιστικός. Σε διαφορετικές συνθήκες είναι πολύ καλύτερο και πιο αποτελεσματικό για την κοινωνία να έχει κάποιο συνεργατική συμπεριφορά. Όμως, για τις ε, προαγωγές ε, άρρητο στοιχείο ε, είναι πάντοτε ο ανταγωνισμός και δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και δεν χρειάζεται να τα συζητήσουμε, να διακόψουμε εδώ τη συζήτηση και να πούμε ότι δεν ισχύει αυτό. Αλλά πραγματικά εγώ δεν ερμηνεύω έτσι την κατάσταση. Ο στόχος της ε, μελέτης ποια ποιος είναι να βρούμε έναν επιπρόσθετο παράγοντα για να δούμε για ποιο λόγο υπάρχουν αυτές οι διαφορές στην αγορά εργασίας. Και όπως σας είπα στα αρχικά μου σχόλια, φυσικά υπάρχουν διαφορές όταν μιλάμε για τη συνεργασία και τα συνεργατικά πρότυπα. Αλλά αυτό δεν ισχύει όταν μιλάμε για την αύξηση μισθού ή για την προαγωγή, για την συμφιλίωση της οικογενειακής και επαγγελματική ζωής και πώς αυτό έχει αρνητικό αντίκτυπο για, την, ε, για το μέλλον ε, κάποιας. Ε, το θέμα θέμα είναι πώς ε, πρέπει να το χειριστούμε. Εγώ δεν διαφωνώ. Είναι καταπληκτικό να συνεργαζόμαστε, αλλά στο κάτω-κάτω της γραφής πώς αλλάζει κάτι που πρέπει να αλλάξει και πώς κάποιοι πρέπει να δέχονται ε, ε, ορισμένες φορές την πρόκληση του ανταγωνισμού. Εντάξει, είναι εύκολο να πείτε ότι εσείς είστε ε, ε άντρες και φυσιολογικό είναι αυτό, αυτό που μας λέτε, αλλά ορισμένες φορές μέσα στη ζωή υπάρχουν ε, συνθήκες οι οποίες καθιστούν απαραίτητο τον ανταγωνισμό. δεν διαφωνούμε, απλώς έχουμε διαφορετική εστίαση. Εγώ στην ε, ομιλία μου ε, θέλησα να εστιάσω σε αυτή τη διάσταση του ζητήματος. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Θα σταματήσουμε εδώ. Θα ε, κλείσει εδώ και αυτός ο γύρος. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές. Θα ήθελα να προσκαλέσω στο βήμα τους ομιλητές για τον επόμενο γύρο. Εδώ μπορούμε να συζητήσουμε για τα διδάγματα, μπορούμε να κλείσουμε από την καταπολέμηση του φαινομένου ανεργίας των νέων, έχοντας υπόψη το πόσο σημαντικό είναι για τους νέους να βρουν ε, μια θέση. Ε, έχουμε και δύο σκιώδεις ηγητές και εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, θα ακούσουμε τη συμβολή τους λοιπόν ε, στο σημερινό σεμινάριο. Θα αρχίσουμε με την κυρία Λιμπεράκη που θα εξετάσει το θέμα ε, των ε, ήδη προταθέντων μέτρων ε, στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως τον αντίκτυπο της εγγύησης για τους νέους και πώς θα επηρεάσει αυτό την είσοδο των νέων στην αγορά εργασίας. Είναι ερευνήτρια στο στην Πάντιο, στην Ελλάδα και ε, ε, έχει δικαιωθεί σε αυτά ε, τα ζητήματα με ευρωπαϊκή προοπτική. Θα σας ακούσουμε λοιπόν ευθύς αμέσως. Ευχαριστώ. Ε, ε, αντιλαμβάνομαι ότι ήταν τόσο ενδιαφέρουσες προηγούμενες παρουσιάσεις που ίσως έχετε υπερφορτιστεί. Εγώ θα ήθελα ε, να σχολιάσω αυτό το πακέτο για τους νέους και κατά πόσο θα βοηθήσει τους νέους και τις νέες για να σωματωθούν στην αγορά εργασίας. Το αναχείριο ζήτημα ποιο είναι ουσιαστικά. Αυτό που θα έπρεπε να μας ε, ανησυχεί και αυτό που όντως φαίνεται να ανησυχεί την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ε, οι σχέσεις των νέων με την κοινωνία που φαίνεται σε διάφορες περιστάσεις να δυσλειτουργούν. Φυσικά, ε, ο αντίκτυπος ε, της ε, κρίσης της απασχόλησης μπορεί να έχει διαφορετικές εκφάνσεις. Όντως έχει σημασία και η ηλικία και το φύλλο και ο κλάδος και η εκπαίδευση που έχει κάποιος. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να γενικεύουμε από τη γενική εικόνα της ε, κρίσης να υποθέσουμε ότι η ανεργία των νέων είναι μια μινιατούρα της ε, συνολικής εικόνας. Ε, αυτό δεν προκύπτει αυτόματα. Ακόμη και ο παράγοντας φύλλο ε, στο φαινόμενο της ανεργίας των νέων ε, μου φαίνεται ότι διαφοροποιείται από τις διαφορές σε πιο προχωρημένες ηλικίες, άνω των 35 για να είμαι πιο συγκεκριμένη. Οι στρατηγικές και οι πολιτικές και τα πακέτα πολιτικών θα πρέπει να συνυπολογίσουν όλες αυτές τις περίπλοκες διαστάσεις του ζητήματος. Επίσης θα πρέπει να συνυπολογίζουν πως οι πολιτικές, ακόμη και όταν δεν είναι πολύ αποτελεσματικές, παρόλα αυτά επηρεάζουν την εικόνα που έχουν οι άνθρωποι για τους ίδιους, τι είδους εναλλακτικές έχουν, και με ποιο τρόπο μπορούν να συνεχίσουν, ε, πώς θα διαμορφωθεί η μελλοντική του συμπεριφορά στην αγορά εργασίας. Είναι σημαντικό λοιπόν να τονίζουμε ε, σε σχέση με αυτά τη διάσταση του φύλου. Όταν εξετάζουμε λοιπόν τα ποσοστά ανεργίας, αυτό που βλέπουμε στην ευρύτερη εικόνα στην Ευρώπη και ε, καταλαβαίνω και συμφωνώ ότι δεν είναι χρήσιμο πάντα να μιλάμε για την Ευρώπη των 25 γιατί υπάρχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά σε ομάδες, σε κρατών κτλ. Αλλά σε δεκάλεπτη παρουσίαση δεν γίνεται να πω σε περισσότερε λεπτό. Η γενική εικόνα ποια είναι λοιπόν ότι αυξήθηκε η ενεργεία των νέων κατά τη διάρκεια της κρίση όλε τι χώρε. Ωραία. Επίσης ενδιαφέρον είναι να δούμε σε χώρες όπου είναι υψηλό ε, το ποσοστό ανεργία, σε χώρες ε, όπου οι οικονομολόγοι και διάφοροι άλλοι μιλάνε για το εθνικό ποσοστό ανεργίας, ε, το μακρο το ποσοστό της μακροχρόνιας ανεργίας σε αυτές τις χώρες ήταν υψηλό πριν την κρίση και όταν συνέβαινε αυτό αυξανόταν ε, και ε, σε απόλυτους και σχετικούς όρους πολύ πιο γρήγορα μετά την κρίση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι νέοι που ζουν σε χώρες όπου ήταν υψηλά τα ποσοστά ανεργίας προ-κρίση είναι ακόμη, σε ακόμη πιο ευάλωτη θέση μετά την κρίση. Ε, δεν υπάρχει διακριτό όμως μοντέλο σε σχέση με τις διαφορές των δύο φίλων ακόμη και σε αυτές τις χώρες. Στην Ελλάδα, Φερρυπίν, είναι συχνότερη απασχόληση των γυναικών ε, παρά των ανδρών κατά 17% είναι υψηλότατο αυτό το ποσοστό. Στην Ισπανία υπάρχει μεγαλύτερη ισορροπία σε σχέση με την ανεργία των νέων. Στην Ιρλανδία βλέπουμε αντίθετες τάσεις σε σχέση με την Ελλάδα. Οι νέοι ε, φαίνεται να είναι σε πιο ευάλωτε σε σχέση με τις γυναίκες. Αυτή η γραφική παράσταση σας δείχνει πράγματα που γνωρίζετε ήδη θέλω να ε, παραμείνουμε σε αυτό. Μόνο να σας πω πως όταν μιλάμε για ποσοστά ανεργία στις τάξεις ε, του 22-23% σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27, οφείλουμε να διαπιστώσουμε ότι είναι πάρα πολύ υψηλό αυτό το ποσοστό. Αυτό το ποσοστό όμως ε, πώς θα ερμηνευθεί είναι λίγο δύσκολο, διότι υπολογίζεται ο αριθμός των νέων που προσπαθούν να απασχοληθούν, όμως ο παρονομαστής του λόγου αυτού είναι ο αριθμός των νέων που με δραστήριο τρόπο μετέχουν στην αγορά εργασίας, είτε επειδή ε, ε, έχουν ήδη μια θέση απασχόληση είτε επειδή δραστήρια αναζητούν μια. Πάνω από 50% των νέων όμως ε, εκφεύγουν του υπολογισμού αυτού για τον υπολογισμό του ποσοστού ανεργίας. Όμως εάν χρησιμοποιήσουμε ένα διαφορετικό παρονομαστή και χρησιμοποιήσουμε όλη την πληθυσμιακή ομάδα ε, από τα 15 έως τα 24 έτη τότε θα έχουμε το ίμιση και αυτό δεν μας ξαφνιάζει διότι οι μισοί νέοι μετέχουν είτε σε ε, κάποια εκπαίδευση ή έχουν κάποια θέση απασχόλησης. Αυτό με φέρνει στο θέμα της, ε, ε, των NEET, των ανενεργών νέων που ούτε απασχολούνται ούτε συμμετέχουν σε κάποια εκπαίδευση στο, στην πληθυσμιακή ομάδα 15-24 χρονών. Εκεί το ποσοστό είναι σαφέστατα χαμηλότερο. Είναι 12,9-13% σχεδόν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι χαμηλότερο το ποσοστό αυτό σε σχέση με το ποσοστό ανεργίας ε, όπως συμβατικά υπολογίζεται για ε, μεγαλύτερες ηλικίε, όμως είναι πολύ υψηλότερο σε σχέση με τον λόγο για που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό τη ανεργία ε, και στον οποίο προαναφέρθηκα, δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε ολόκληρο τον πληθυσμό ω παρονομαστή σε αυτό το λόγο. Τι είναι ενδιαφέρον σε αυτό αυτήν την κατηγοριοποίηση, σε αυτή την ε, έννοια. Ε, θα πρέπει κάποιος να ασχοληθεί όχι μόνο με τα όσα συμβαίνουν ε, στους νέους ε, που με δραστήριο τρόπο αναζητούν θέση απασχόλησης, αλλά το τι συμβαίνει γενικότερα στους νέους και οι συζητήσεις που γίνονται σε σχέση με την έννοια του NEET, ε, του ανενεργού νέου, τονίζουν το σύνολο αυτής της πληθυσμιακής ομάδας και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Όταν λοιπόν κάποιος εξετάζει αυτή την πληθυσμιακή ομάδα που ε, ε, ε, των ανενεργών νέων δεν έχουν θέση απασχόληση, δεν καταρτίζονται, δεν μετέχουν σε καμία μορφή εκπαίδευση, οι NITS. Είναι δύσκολο να έχουμε ένα διακριτό, ξαναλέω, μοντέλο σε σχέση με τη διαφορά των φίλων Υπάρχει όμως ένα στοιχείο, τουλάχιστον ένα, που, στο οποίο αναφέρθηκε ο πρώτος ομιλητή όταν ερωτήθηκαν ε, κάποιοι νέοι για ποιο λόγο δεν απασχολούνται ή δεν ε, αναζητούν μια θέση απασχόλησης, ε, η συνήθιση ύποπτη είναι κάποια αναπηρία ή κάποια ασθένεια και φαίνεται ότι είναι συχνότερο αυτό στους νέους παρά στις νέες. Ε, οι οικογενειακές ευθύνες, όχι όμως η περίθαλψη κάποιου οικογενειακού μέλους, ε, για τις νέες ε, ε, είναι πολύ σημαντικός παράγοντας, 16,3% για τις γυναίκες έναντι 10,6% για τους άντρες. Όμως και πάλι η διαφορά δεν είναι τόσο σημαντική. Εκεί που εντοπίζεται μια όντω αισθητή διαφορά είναι στον τομέα της περίθαλψης των παιδιών ή των ηλικιωμένων ή των ε, αναπήρων μελών της οικογένειας. Οι νέες ε, που εντάσσονται στην ομάδα ΝΙΤΑ αυτή την απάντηση δίνουν ε, και το ποσοστό είναι 35,3% των ερωτηθήσεων. Επίσης, είναι σημαντικό το ότι οι νέοι αποθαρρύνονται περισσότερο, δηλαδή δεν ψάχνουν δουλειά διότι θεωρούν ότι δεν υπάρχει δουλειά. Ενώ οι νέες ε, το ανέφεραν ε, σε λιγότερο από το ίμιση των περιπτώσεων ως πιθανή αιτία. Αναρωτιέμαι λοιπόν ποιες είναι οι αιτίες, ποιοι είναι οι παράγοντες ε, που έχουν ε, μεγαλύτερη σημασία ε, για να οδηγήσουν ε, νέους να γίνουν νίτ, ανενεργοί. Ξέρουμε στην περίπτωση αναπηριών ότι οι νέοι που πάσχουν έχουν 40% περισσότερες πιθανότητες να εισέλθουν σε αυτή την κατηγορία. Υπόβαθρο μεταναστευτικό 70% περισσότερες πιθανότητες ε, και είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να το λάβει σοβαρά υπόψη αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες η χαμηλή μόρφωση ε, όταν προέρχονται από μακρισμένες περιοχές ή από οικογένειες χαμηλού εισοδήματος. Αυτοί είναι οι βασικοί ε, παράγοντες ε, που σπρώχνουν τους νέους ε, προς αυτήν την κατηγορία ανεξαρτήτως κρίσης. Με την κρίση προστίθενται και άλλοι δύο παράγοντες κινδύνους. Οι χώρες που εκτίθενται σε ακραίες μορφές αυτής της κρίσης, όπως φαντάζεστε, έχουν την πρώτη θέση. Και τώρα να κάνω μια δεύτερη, ένα σχόλιο για ε, για τη δεύτερη κατηγορία ε, οι χώρες με ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς ε, και όσοι έρχονται από τέτοιες χώρες ξέρουν για τι πράγμα μιλώ και εγώ η ίδια εξάλλου οι νέοι προστατεύονται περισσότερο από τις οικογένειες αυτές τις χώρες και αυτό αληθεύει δηλαδή οι γονείς θεωρούν ότι έχουν μία ένα υποχρέωση ανεξαρτήτως ηλικίας να προστατεύουν τα παιδιά τους και ε, τα παιδιά ποτέ δεν γερνάνε σε αυτές τις χώρες στα μάτια των ε, γονιών. Πέρα από αυτήν την ε, προστατευτική ομπρέλα, αυτό καθιστά ιδιαίτερη δυσχερή την πρόσβαση στην ενηλικίωση. Είναι παρατεταμένη, εξαιρετικά παρατεταμένη η διαδικασία της ορίμανσης σε περίοδο υψηλής ανεργίας και υψηλής ανασφάλειας. Αυτό θα είναι το χειρότερο που μπορεί να κάνει κανείς ε, στο παιδί του, να μην το επιτρέπει με αυτή τη συμπεριφορά να ρισκάρει. Ε, λοιπόν, είμαι σε μια χώρα που είναι ε, σοβαρότατα εκτεθειμένη στην κρίση, αλλά όπου ταυτόχρονα είναι ισχυρότατη η οικογενειακή δεσμή, εάν συνδέαστε τους δύο παράγοντες, είναι καταδικασμένη η χώρα. Η οικονομική θεωρία μας μαθαίνει ότι όταν είναι υψηλή ενεργεία και ε, ε, κρίση οικονομική, ε, δύο είναι οι πιθανές αντιδράσεις των νέων. Είτε αποθαρρύνονται και λένε «Α, δεν υπάρχει δουλειά, οπότε τι να κουράζομαι, δεν υπάρχει δουλειά» και αποσύρονται από την αγορά εργασίας, το εφέ του αποθαρρυμένου εργαζόμενου ή κάποιοι άλλοι επειδή ε, έχουν εξορθολογήσει τον τρόπο σκέψης τους, ε, ε, πιστεύουν ότι για να συντηρήσω την οικογένειά μου ή τις δικές μου συνθήκες διαβίωσης, θα δραστηριοποιηθώ περισσότερο στην εξέβρεση μιας θέσης απασχόλησης. Λοιπόν, για το σύνολο του εργατικού δυναμικού φαίνεται ότι ε, οι γυναίκες ε, είναι πολύ πιο δραστηριές στη δεύτερη κατηγορία, ε, κυρίως σε περίοδο κρίσης παρά σε αυτή την κατηγορία των αποθαρρυμένων εργαζομένων. Όμως αυτό δεν ισχύει για νέους κάτω από 25 χρονών. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Τι, γιατί σημαίνει στις γυναίκες πάνω από το, άνω των 25 ε, για να δείχνουν αυτήν την αιμονή και την αποφασιστικότητα να ε, προσπαθούν να ε, βρούνε μία θέση απασχόλησης ε, ενώ έχουν εισέλθει στην κατηγορία των ανέργων που λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας το οποίο είναι χαμηλό στη συγκεκριμένη περίπτωση σε σχέση με τους άντρες που άνω των 25. Και γιατί κάτω από το ε, κατόφλι των 25 ε, τα δύο φύλλα υιοθετούν την ίδια στάση που ε, φαίνεται να τους οθεί προς την πρώτη κατηγορία του αποθαρρυμένου εργαζόμενου. Αυτό που ξέρουμε από προηγούμενες έρευνες ε, για τις πρακτικές ασκήσεις και το πώς επηρεάζει το φύλλο αυτές, ε, οι εργοδότες όταν έχουν έλλειψη δεξιοτήτων ε, τείνουν να προσλαμβάνουν τέτοιους εργαζόμενους. Επίσης, η κατάρτιση όταν ενέχει διακριτικές μεταχειρήσεις είναι, μπορεί να συγκριθεί με τις διακριτικές μεταχειρήσεις ε, που παρατηρούνται στην αγορά εργασίας ε, και έχουμε έτσι χαμηλόμιστες θέσεις εργασίας και αντίστοιχα ε, οι πρακτικές ασκήσεις για τις γυναίκες διαρκούν λιγότερο και αμείβονται λιγότερο επίσης. Αυτό αντανακλάται στις μισθολογικές διαφορές και στον επιμορισμό των θέσεων εργασίας ανάμεσα στα δύο φύλλα. Ε, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την, ε, ε, την κατάσταση ως προς αυτές τις ε, διαφορές. Το πρώτο που μπορούμε να κάνουμε είναι να καταπολύσουμε το φαινόμενο στην αγορά εργασίας, στην κατάρτιση και το πεδίο της πρακτικής άσκησης είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έγιναν πειράματα που έδειξαν ότι οι καθηγητές μπορούν, ενδέχεται να μεταχειριστούν διαφορετικά τα δύο φύλλα, ακόμη και σε πολύ μικρές ηλικίε, όταν διδάσκουν μαθηματικά, διότι προσμένουν διαφορετικές επιδόσεις. Βλέπουμε λοιπόν τα τρία αγόρια που φαίνεται να είναι πολύ δραστήρια. Όλοι οι υπόλοιποι ροχαλίζουν στο μάθημα διότι... Ε, και έχουμε την εντύπωση ότι Πρόκειται για μια ε, διακριτική μεταχείριση, η οποία όμως δεν αντανακλάται στα στατιστικά στοιχεία, διότι συμβαίνει μέσα στο μυαλό των δασκάλων ή των καθηγητών και ε, διαχέεται και στα ε, μυαλά των μαθητών ή των φοιτητών. Πρόκειται για λιγότερο ορατές μορφές διακριτικής μεταχείρισης. Ε, φαίνεται ότι οι μεγάλοι εργοδότες ε, είναι πιο ανοιχτοί ως προς την ε, εξή ιδέα. Να προκρίνουν την καλύτερη κάλυψη των αναγκών των δύο φύλων ως προς τις πρακτικές ασκήσεις και αυτό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για μελλοντικές πολιτικές. Κάτι άλλο που είναι σημαντικό. Εάν στην οικογένεια του νέου υπάρχει κάποιος που έχει άτυπη μορφή εργασίας ή που έχει επιλέξει μια άτυπη μορφή εργασίας ε, ως προς τα στερεότυπα των δύο φίλων. Εάν η μητέρα είναι αστροναύτης, παραδείγματος χάρη, τότε οι νέοι τείνουν περισσότερο να επιλέξουν ε, μη τυπικές για το φύλλο τους ε, πρακτικές ασκήσεις. Ε, με την κρίση μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση ως προς την πρακτική άσκηση και ε, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το στοιχείο. Ε, στην εκπαίδευση όμως ε, ε, βασικά είναι που πρέπει να ενσωματώσουμε τον παράγοντα φύλλο και μιλώντας για την εκπαίδευση θα πρέπει να καλύψουμε και τα νηπιαγωγεία διότι θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το τι συμβαίνει στο, σε αυτή τη μικρή ηλικία. Μπορώ να συνεχίσω. Ένα λεπτάκι, ωραία το πακέτο για τους ε, νέους θα πρέπει να ενέχει όλε αυτές τις ε, προτεραιότητε, να συνυπολογίζει το παράγοντας φύλλο, αλλά είναι κρίμα το εξή. Παρότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μία σειρά από πολιτικές ε, για να προωθεί την ισότητα των δύο φύλων και ασχολείται με αυτό το ζήτημα και ε, την αντιμετώπιση του προβλήματος. Μέσα στο πακέτο για τις εγγυήσει των νέων δεν αναφέρεται καθόλου ε, ο παράγοντας φύλλο, κάτι που ξαφνιάζει. Ε, η φραζολογία και ο σχεδιασμός του ίδιου του πακέτου ίσως δεν εξυπηρετούν το στόχο της ε, κατάργησης των διαφορών, της καταπολέμησης μάλλον των διαφορών ανάμεσα στα δύο φύλλα. Ε, η αποτίμηση πρέπει να γίνεται σε όλα αυτά τα επίπεδα κατά το σχεδιασμό του πακέτου και τα ζητήματα φύλου πρέπει επίσης να ε, συνυπολογίζονται όταν επεξεργαζόμαστε το σύστημα ποιοτική αξιολόγηση για τις πρακτικές ασκήσεις. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντική ανταλλαγή των βελτίστων πρακτικών τον τομέα των μη τυπικών πρακτικών ασκήσεων, να κινητοποιήσουμε όποια θετική εμπειρία έχουμε, πρέπει να την προωθήσουμε και να ε, την καταστήσουμε υποδειγματική. Ε, και τέλος, Αλεξίου, σημαντικό θα ήταν να πούμε ότι ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να αποδοθεί ε, στην κατάσταση των νέων που φροντίζουν μέλη της ε, ε, οικογένειας. Οι νέοι ε, μπορεί να έχουν πολύ περισσότερες διαφορές συμπεριφορά τους σε σχέση με αυτά που πιστεύουμε συγκρίση με πιο ηλικιωμένους συγγενείς τους. Πρέπει να σκεφτόμαστε ταχύτερα και να δρούμε ταχύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Δηλαδή γνωρίζουμε ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των φύλων όταν αποθαρρύνονται αλλά εν γέννη αλλά όχι όσον αφορά τους νέους. Ευχαριστώ για μία ακόμη φορά, ευχαριστώ πολύ. Έχουμε χρόνο για ερωτήσεις αργότερα. Προχωράμε στον επόμενο μιλητή, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η κυρία Νταουάν επεξεργάζεται μελέτη που σχετίζεται με την ανεργία των νέων. Ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συνεδρίαση και ευχαριστώ που μου δίνει την ευκαιρία να πάρω το λόγο εκπροσωπώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θα αναφερθώ ξανά στα στοιχεία και στις έρευνες ε, που συζητήθηκαν και σχολιάστηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίασης και που δίνουν σε εκείνους που αποφασίζουν σε πολιτικό επίπεδο δυνατότητα δράσης και αντίδρασης όπως τα αποτελέσματα όσον αφορά της πειραματικής οικονομίας που είναι πολύ υπέρ των ποσοστώσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν χρειάζεται να πιστεί επί των ποσοστώσεων διότι η Επίτροπος Vivian Ρέντινγκ έχει προτείνει ποσοστώσεις τον περασμένο Νοέμβριο αλλά τώρα το θέμα είναι στα χέρια των δύο συνομοθετών και είμαι βέβαιη ότι τα αποτελέσματα που ανακαλύψαμε σήμερα μπορεί να είναι πολύ χρήσιμα στις συζητήσεις. Αυτό που θα κάνω θα είναι να παρουσιάσω τις δρομολογηθήσεις δράσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο που τείνουν να απαντήσουν στα προβλήματα που αναφέρθηκαν σήμερα που είναι ταυτόχρονα προβλήματα συγκυριακά διότι η ανεργία των νέων είναι πολύ ευαίσθητη έναντι της οικονομικής συγκυρίας. Η ανεργία των νέων είναι πολύ ψηλή διότι υπάρχει μια έλλειψη θέσεων απασχόλησης, αλλά είναι και αυτό που συζητήσαμε σήμερα ουσιαστικά. Υπάρχουν προβλήματα πιο διαθροτικά που συνδέονται με τις ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών. Για να παρουσιάσω λοιπόν τις πολιτικές που έχουν δρομολογηθεί σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, θα αναφέρω τέσσερα σημεία Τη δημόσια Υπηρεσία απασχόληση, προ επαγγελματικού προσανατολισμού και τα θέματα τη παιδεία. Η προηγούμενη ομιλήτρια ανέφερε σε ποιο βαθμό η καταπολέμηση των στερεοτύπων εντό των υπηρεσίων παιδεία ήταν κάτι σημαντικό και αυτό ήθελα να συζητήσω. Σε δεύτερο σημείο θα αναφερθώ σε θέματα συμφιλίωση και δύο τελευταία σημεία θα είναι περισσότερο προβληματισμοί και σκέψει διαδικαστικού τύπου όσον αφορά τις συνεργασίες και συμπράξεις και τη χρηματοδότηση. Λοιπόν, πρώτο σημείο να επενθυμίσω ότι το πακέτο για την απασχόληση των νέων, το οποίο θετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τέλος ε, του 2012, ε, αναγνώριζε τις ανισότητες που υπήρχαν μεταξύ ανδρών και γυναικών σε ζητήματα που άπτονται της αγοράς εργασίας κυρίως όσον αφορά τους νέους άνδρες και τις νέες γυναίκες και ότι το βασικό στοιχείο του πακέτου για την απασχόληση που είναι μια σύσταση προς τα κράτη-μέλη να θεσπίσουν εγγυήσει για τους νέους, ζητά από τα κράτη-μέλη να λάβουν υπόψη τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στους νέους και τις διαφορές που υπάρχουν ε, όσον αφορά τα φύλλα. Αυτή η πρόταση συμπεριλήφθη πλήρως από το Συμβούλιο, την ενέκρινε και οθέτησε τη σύσταση που αφορά την εγγύηση για την απασχόληση που πρέπει τώρα να εφαρμοστεί επιτόπου ουσιαστικά από τις δημόσιες υπηρεσίες της αρμόδιας για την απασχόληση. Οι υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού ανάντι στον τομέα της παιδείας ε, έχουν ένα ρόλο να παίξουν. Ε, διοργανώσαμε μια ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών όπως αποκαλείται με τα κράτη-μέλη στο τι μπορούμε να κάνουμε σε επίπεδο προσανατολισμού πολύ νωρίς στα πλαίσια του εκπαιδευτικού συστήματος. Ε, ξέρετε, στη Γερμανία, παραδείγματο χάρη, υπάρχει το Boys Day και Girls Day, οι μερίδες αγοριών και κοριτσιών, όπου δείχνουν εκεί στα νέα κορίτσια ποια επαγγέλματα μπορούν να ακολουθήσουν τον τεχνικό τομέα και ποια είναι τα επαγγέλματα στον τομέα του care, ε, της φροντίδας στα νέα αγόρια. Ε, το εξετάσαμε το θέμα και έγινε προβληματισμό στα κράτη-μέλη. Πρόσφατα, το περασμένο φθινόπωρο, έγινε μια ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών και προβληματισμό όσον αφορά την εξάλληψη των στερεοτύπων όσον αφορά ε, τα εγχειρίδια, τα σχολικά και το πρόγραμμα σχολικών μαθημάτων. Παίρνω παραδείγματα από τη Δανία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και η Γαλλία ενδιαφέρεται για αυτά τα ζητήματα. Αναφέρονται αυτά τα θέματα στον τύπο. Το βασικό μήνυμα που συγκρατώ είναι ότι στα κράτη-μέλη υπάρχουν πολλές πρακτικές που φαίνονται ενδιαφέρουσες, που δεν έχουν αξιολογηθεί πλήρως, αλλά αποπειρώνται να καταπολεμήσουν τα στερεότυπα και τον διαχωρισμό των φύλων στην αγορά εργασίας, ακόμα και αν τα στοιχεία παραμένουν σχετικά σταθερά στον τομέα. Θα ήθελα να προσθέσω επίσης ότι ευρωπαϊκά ταμεία είναι πάρα πολύ χρήσιμα σε αυτό το τομέα, ευρωπαϊκή πόρη, συζήτησα πέρσι με το διευθυντή του UNICEF που είναι το κέντρο προσανατολισμού το γαλλικό που μου έλεγε ότι χάρη στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μπόρεσε να πραγματοποιήσει μια εκστρατεία ευαισθητοποίηση των νέων κοριτσιών και των νέων αγοριών όσον αφορά την καταπολέμηση των στερεοτύπων. Κατέληξα με το πρώτο σημείο. Το δεύτερο μου σημείο αφορά την συμφιλίωση αυτή που αναφέραμε μέσω των διαφόρων παρουσιάσεων Σήμερα είδαμε σε ποιο βαθμό ήταν ο γόρδιος δεσμός του προβλήματος των ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί αυτό το θέμα εκ του σύνεγγυς. Κυρίως παρακολουθεί την εφαρμογή των στόχων της Βαρκελόνης όπως αποκαλούνται. Το 2002 δεσμεύτηκαν τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν τις υπηρεσίες αποδοχής ε, και μέρημνες των μικρών παιδιών, ούτως ώστε τα παιδιά που είναι κάτω από τριών ετών, 33% των παιδιών κάτω από τριών ετών να μπορούν να δέχονται αυτή τη μέρημνα στις επίσημες υπηρεσίες και οι 90% των παιδιών από τρία μέχρι την υποχρεωτική, με την ηλικία υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων να παρακολουθούνται από τις επίσημες υπηρεσίες, να φροντίζονται στις επίσημες υπηρεσίες. Το 2010 ε, είπαμε ότι θα δημοσιεύσουμε και δημοσιεύσουμε σύντομα μία έκθεση σχετικά με αυτούς τους στόχους. Μπορώ να σας αποκαλύψω κάποια στοιχεία. Ε, δημοσιεύτηκαν τα στοιχεία από τη Eurostat ε, πρόσφατα. Οι στόχοι δεν θα επιτευχθούν. Όμως βλέπουμε μία βελτίωση των επιδόσεων όσον αφορά τις υπηρεσίες υποδοχής των μικρών παιδιών. Για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ισχύει αυτό. Όμως ε, υπάρχει μία μείωση όσον αφορά το ποσοστό της κάλυψης σε κάποιες χώρες τα τελευταία δύο χρόνια. Και εκεί τα διευθυντικά ταμεία είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Υπάρχουν χώρες όπως είναι η Πολωνία, η Ουγγαρία που χρησιμοποιούν μαζικά τα διευθυντικά ταμεία για να αναπτύξουν αυτές τις υπηρεσίες μέρημνας για τα μικρά παιδιά. Μου μένουν μερικά λεπτά για να σας ε, μιλήσω για τη χρηματοδότηση για όλες αυτές τις δράσεις. Ε, πιστεύω ότι το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έστειλε ισχυρό μήνυμα θέλοντας να κινητοποιήσει ένα μέρος των πόρων για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων ε, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από αυτό είχε επεξεργαστεί πριν την κρίση το θέμα της κινητοποίησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και παρουσίασε τον Μάρτιο, τον περασμένο Μάρτιο μια αξιολόγηση της κινητοποίησης των διαθωτικών ταμείων για την καταπολέμηση της ανεργία των νέων και τελευταίο μου σημείο θα αφορά τα διαδικαστικά θέματα και τις συμπράξεις εταιρικέ σχέσεις. Λέγαμε σήμερα το πρωί στη συνεδρίαση της Επιτροπής σε ποιο βαθμό έπρεπε όλες αυτές οι πολιτικές να ασκούνται μαζί με τους νέους Υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο το Ευρωπαϊκό Φόρουμ των Νέων που είναι μια επικοδομητική φωνή και ενεργή φωνή που εκπροσωπεί τους νέους και είναι πάρα πολύ χρήσιμο ότι την ακούει κανείς και όλα αυτά τα μέτρα της κατάρτισης για την καταπολέμηση ανεργίας δεν μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς τους κοινωνικούς εταίρους. Επί παραδείγματι διαβολευτήκαμε τους κοινωνικούς εταίρους για την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού πλαίσιου ποιότητας όσον αφορά τις μαθητείες και την ε, κατάρτιση και μετά από αυτές τις διαβουλεύσεις θα παρουσιάσουμε ε, το πλαίσιο αυτό που σας προανέφεραν. Κατά κλειδί θα έλεγα απλώς ότι αυτά που ανέφερα είναι λεπτομερέστερα στην ετήσια έκθεση που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε στις 8, θα δημοσίευσε στις 8 Μαΐου για την ενισότητα μεταξύ ανδρών και νεγών. Θα βρείτε και παραδείγματα βελτίστων πρακτικών σε εθνικό επίπεδο. Η σημαντικότερη εξέλιξη οι σημαντικότερε εξελίξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, και οι διάφοροι δείκτες κλειδιά στου διάφορου τομεί αναφέρονται. Ευχαριστώ για την προσοχή σα. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ εκ νέου ε, που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπόρεσε να παρίστα τι εργασίε. Ευχαριστώ πάρα πολύ ε, για την παρέμβασή σα και μπορούμε να προχωρήσουμε και να πάμε στον επόμενο μιλητή. Η κυρία Φλάβια Πέσκε που έκαθιστε εκεί από το IRS και θα έχετε ενδιαφέρον καθήκον να συναγάγετε κάποια συμπεράσματα από αυτή την ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Δεν σας ζηλεύω. Είσαστε η τελευταία που θα πάρετε το λόγο και θα πρέπει να συναγάγετε τα συμπεράσματα. Όλοι έχετε δοκτορά, έχετε δοκτορά στις κοινωνιολογικές επιστήμες εργαστήκατε σαν ελεύθερη επαγγελματία από το 1993 και από το 1999 είστε ανώτερη ερευνήτρια όσον αφορά τη μονάδα για τις εργασιακές πολιτικές και ασχολείστε με τα θέματα τη συμπερίληψη των θεμάτων όπως φίλου στι διάφορε πολιτικέ που ασκούνται και είστε ειδικοί για τι πολιτικέ, για την ισότητα των φίλων, για την κοινωνική ένταξη, για πολιτικέ αγορά-εργασία και τα διάφορα συναφή θέματα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω Ιταλιστή που είναι η μητρική μου γλώσσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση και όπως είπε και ο κύριος Γκούσταυσον έχω τη δύσκολη αυτή θέση να είμαι η τελευταία που παίρνει το λόγο σε αυτό το απόγευμα και να μπορέσω να συναγάγω τα συμπεράσματα από όλες τις πτυχές που αναφέρθηκαν σήμερα. Θα προσπαθήσω συνεπώς να ακολουθήσω εν μέρη το σημείωμα που ετοιμάστηκε και που έχετε στα, στο, στα έγγραφά σας και να συνοψίσω αυτά που ανέφεραν οι εμπειρογνώμονες στις διάφορες παρουσιάσεις που προηγήθηκαν. Ε, σίγουρα ε, είδαμε από τις προηγούμενες παρουσιάσεις πως το θέμα της ανεργίας των νέων συνδέεται στενά με τις διάφορες με τη μετάβαση από το σχολείο στην εργασία, διάφορε μορφέ διακρίσει και με διάφορα φαινόμενα διαθωτικά που επηρεάζουν με διαφορετικό τρόπο την ομάδα στόχο των νέων, όπως αποκαλείται. Χωρίς να εισάγουμε τη μεταβλητή του φίλου, σίγουρα αυτή η ομάδα δεν είναι ομοιογενής και απαιτεί λοιπόν να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες και διαφορές ε, που βρίσκονται εντός των νέων. Υπάρχουν υποομάδες πιο ευάλωτες που πρέπει να αντιμετωπίσουν δυσχέρειες στο να μπορέσουν να εισέλθουν και να παραμείνουν στην αγορά εργασίας. Αυτό προφανώς εδώ πρέπει να εξετάσουμε αυτές τις πτυχές ε, υπό την έποψη και των φίλων. αν βάλουμε και τη συνιστόσα των φίλων μέσα, περιπλέκεται η εξίσωση. Όσον αφορά, τους, αν λάβουμε υπόψη πέρα από τους νέους σας σύνολο και τις ε, νέες κοπέλες και τα νέα αγόρια, οι παρεμβάσεις που έγιναν σήμερα, ε, περιέχουν αυτό το στοιχείο. Που είναι και το κρίσιμο στοιχείο θα έλεγα. Και μετά πρέπει να μπορέσουμε να καταφέρουμε να εφαρμόσουμε πολιτικές και μέσα και εργαλεία και παρεμβάσεις που θα καθορίζονται επί τη βάση των ιδιαίτερων αναγκών κάθε νέου αγοριού και νέας κοπέλας. Τονίστηκε η σημασία που, έχει μία ανάλυση που πρέπει να διεξαχθεί με βάση το φύλλο και όσον αφορά την άλυση των στοιχείων και των φαινομένων που χαρακτηρίζουν τη διάσταση της απασχόλησης και της ανεργίας των νέων και όσον αφορά την ανάλυση των πολιτικών και των παρεμβάσεων που θα μπορέσουν να δρομολογηθούν. Εντάχει θα αναφερθώ σε κάποια παραδείγματα που βρίσκεται και στο σημείωμα και που αναφέρθηκαν και στις προηγούμενες παρεμβάσεις. Διεφάνει και είναι σαφές αυτό ότι πάρα πολλά από τα φαινόμενα που συνήθως συνδέονται με την απασχόληση και την ανεργία των νέων τα θέματα αυτά αντιμετωπίζονται ουδέτερα χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές των φύλων και όλες αυτές οι αναλύσεις εμφανίζονται μια στιγμή όπου χρειάζεται διαφορετική προσέγγιση. Να διαβάνεται υπόψη η διάσταση του φύλου για να ερμηνευτούν τα φαινόμενα διαφορετικό τρόπο. Όλα αυτά καταδεικνύουν ότι δεν μπορεί να γίνει μια δεν διαφαίνονται αυτά σε μια ουδέτερη ανάλυση και πρέπει αυτά τα φαινόμενα να λυθούν περαιτέρω και δεν αναφέρονται μέχρι τώρα και να αναλύουν τι πολιτικέ που ακολουθούνται και τι παρεμβάσει. Όλοι οι προλαλήσαντε αναφέρθηκαν σε ένα φαινόμενο που αφορά του νετ, δηλαδή αυτού του νέου άντρε και γυναίκε που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Την άκρο ιδιαίτερη. Δεν έχουν ενταχθεί ούτε στον κόσμο της εργασίας, ούτε στον κόσμο της παιδείας και της κατάρτισης ήδη από την πρώτη πρώτη παρουσίαση αναφέρθηκε ότι αν αναλύσει κανείς αυτό το φαινόμενο μέσω μιας προσέγγισης των φίλων η διαφορά μεταξύ νέων ανδρών και νέων γυναικών φαίνεται άμεσα. Το να μιλήσουμε για νετ με έναν τρόπο ακαθόριστο χωρίς να δούμε ακριβώς ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες των νέων ε, ανδρών και νέων νετ γυναικών εκ των πραγμάτων εξουδετερώνει ή καθιστά λιγότερο αποτελεσματικές τις πολιτικές και παρεμβάσεις. Είδαμε ότι οι γυναίκες παραμένουν επί πιο μακρόν παγιδευμένες σε αυτή την κατάσταση και ότι το στάτους τους της αδρανίας ε, είναι σε πιο ψηλό επίπεδο, πιο πολύ πιο μεγάλο από το επίπεδο της αποθάρρυνσης. Αυξάνεται περισσότερο από το επίπεδο της αποθάρρυνσης. Ένα άλλο φαινόμενο όπου γίνεται πιο έντονο αν βάλουμε την συνθήκη, ε, τον όρο της διαφοράς του φύλου από ότι μία, μέσω μίσου ανάλυσης είναι η αλλαγή της κατάστασης όσον αφορά την απασχόληση και την κατάσταση την εργασιακή στην περίοδο της κρίσης αλλά και από την αρχή. Κάτι που χαρακτήριζε ευθύ εξ αρχής την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας αυτή η διαφοροποίηση. Η αύξηση των μορφών ευελιξίας όσον αφορά την εργασία. Και σε αυτή την περίπτωση, εκεί που χρησιμοποιείται μια προσέγγιση που είναι ευαίσθητη στο φύλλο, μπορεί να αναδείξει ότι πολύ συχνά υπάρχει στενή διασύνδεση μεταξύ μορφών πρόσκαιρης απασχόλησης που πλήττουν περισσότερο τις νέες γυναίκες από ότι τους νέους άντρες. Πολλές είναι οι μελέτες που καθορίζουν μια πολύ, πολύ μεγάλο συσχετισμό μεταξύ του γυναικείου φύλου και τις μορφές πρόσκαιρης απασχόλησης που δυστυχώς είναι μια πολύ διαδεδομένη απασχόληση στις αγορές εργασίας των διαφόρων χωρών μελών. Μιλήσαμε σε πολλές παρουσιάσεις που έγιναν, σχεδόν όλοι αναφέρθηκαν στο θέμα της παιδείας, της κατάρτισης, στο επίπεδο της παιδείας και σε αυτή την περίπτωση, χωρίς να λάβουμε υπόψη την προσέγγιση με βάση το φύλλο, μπορούν σχεδόν να έχουμε λαθασμένη εικόνα. Να τυφλωθούμε τους υπήντους εισαγωγικών. Να βλέπουμε την κατάσταση πολύ θετική και να μην είναι. Δηλαδή η δεύτερη παρουσίαση υπογράμμισε πολύ καλά αυτές τις πτυχές. Οι νέες γυναίκες πιο συγκεκριμένα τα τελευταία χρόνια έκαναν βήματα γιγαντιαία ε, αυξήθηκε πολύ σημαντικό αριθμός των νέων γυναικών που έχουν ανώτερη τριτοβάθμια παιδεία που πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο. Και αυτό το φαινόμενο όμως αν ιδωθεί από μια οπτική γωνία με βάση το φύλλο μπορεί να αναδείξει διάφορους άλλους παράγοντες που διαφορετικά δεν θα εμφανιζόταν και δεν θα είχαν αντιμετωπιστεί συνεπώς ανησυχεί τάση μιας ανεργίας μεταξύ των νέων γυναικών που είναι πιο καλά εκπαιδευμένες, με περισσότερα προσόντα, που έχουν μεγαλύτερες δυσκολίες να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, μεγαλύτερη διάρκεια της μετάβασης από το σχολείο στην δουλειά, μεγαλύτερη παρουσία στην άτυπη οικονομία ή σε ευέλικτες μορφές εργασίας, που μπορούν και τείνουν να γίνουν πρόσκαιρες μορφές εργασίας όπως έλεγα. Αυτό μας οδηγεί στο να δούμε στενό συσχετισμό με τον διαχωρισμό όσον αφορά τα σχολικά προγράμματα και την κατάρτιση και όσον αφορά τη διαδρομή από το σχολείο προς τη δουλειά που είναι κρίσιμη σημασία για τους νέους και σε αυτή την περίπτωση αναφέρομαι και σε αυτό που αναφέρθηκε στην τελευταία παρουσίαση, στην παρέμφαση της εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα. Αναφέρθηκε σε όλες τι παρεμβάσεις, σε όλες τι πολιτικές που α, σχετίζονται με τη μαθητεία. Ε, όλα αυτά τα παραδείγματα συνοψίζω. Συνοψίζω για να επαναλάβω και πτυχέ, οι οποίε ήδη προφανώ ήδη αναφέρθηκαν. Όλα αυτά δείχνουν όμω σίγουρα πώς μια προσέγγιση με βάση το φύλλο και συνάδελφος προηγήθηκε πριν αναφέρθηκε ε, στην, ε, στο φορέα αξιολόγηση Συνεπιών... Θα πρέπει να αξιολογηθούν οι συνέπειες, δηλαδή να δούμε πώς μία πολιτική, ένα εργαλείο, μία παρέμβαση μπορούν να έχουν αντίχτυπο διαφορετικό στις γυναίκες και στους άντρες, στους νέους άντρες και νέες γυναίκες. Αυτό είναι σημαντικό στοιχείο. Αν θέλουμε να προγραμματίσουμε πολιτικές και να τις εφαρμόσουμε και να δρομολογήσουμε δράσεις θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις διαφορές που υπάρχουν. Όπως έλεγα στην αρχή, το blindness, η τυφλότης, ε, το blindness όπως στα αγγλικά όσον αφορά το φύλλο, μπορεί να οδηγήσει σε πολιτικέ παρεμβάσει που έχουν τελικά συνέπειε που έχουν τελώ διαφορετικέ από τον αρχικό σκοπό. Δηλαδή, αν δεν λάβουμε υπόψη το... τη διάσταση του φύλου. Διαφορετικό στόχο να πετύχουμε από ότι είχε βά... Ε, στην υπόψη το νομοθέτη. Θα έσβησε κάποια νομοθεσία και κάποια επίδραση, κάποια δράση. Στην παρέμβαση τη συναδέλφου τη Ευρωπαϊκή Επίτροπή, είδαμε ότι υπογραμμίστηκαν οι πτυχέ που σχετίζονται ε, με τις πολιτικές που δρομολογούνται κυρίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να υπάρξει αντίσταση όσον αφορά το φαινόμενο της ανεργίας των νέων. Να καταπολεθεί το φαινόμενο. Όλα τα πακέτα, τα σχετικά, όλες οι δραστηριότητε που έχουν στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων αληθεύει ότι υπάρχουν πάρα πολλά κράτη-μέλη υπό την παρένεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των οργανωμένων ε, φορέων, διαφόρων ενώσεων που ασχολούνται με τα δικαιώματα των γυναικών. Τα κράτη-μέλη έκαναν πολλά πράγματα λοιπόν υπό την πίεση. Κινητοποιήθηκαν διάφορες καλές πρακτικές και πρωτοβουλίες. Αληθεύει επίσης ότι η πτυχή του φύλου εντός πολλών πακέτων νομοθετικών και προτάσεων και δραστηριοτήτων που ενεργοποιούνται σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Η διάσταση του φίλου έλεγα λαμβάνεται υπόψη αλλά όχι τόσο επίσημα. Δεν λαμβάνεται υπόψη ο αντίχτυπος, ο διαφορετικός αντίχτυπος που μπορεί να έχουν οι διάφορες πολιτικές και παρεμβάσεις. Επιδράσεις στους νέους άντρες και νέες γυναίκες. Παράδειγμα, όλες οι πολιτικές και τα μέτρα που έχουν σαν σκοπό να διευκολύνουν τη μετάβαση από τη σχολική ζωή στην εργασία και την πρώτη είσοδο των νέων ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασία. Αναφέρομαι λοιπόν στο πακέτο των μέτρων που αφορούν τη μαθητεία τη εισόδου στην αγορά εργασία που προωθούνται σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Πολύ αυτά τα μέτρα. Θα έπρεπε και σε αυτή την περίπτωση όλα αυτά να διερευνηθούν περαιτέρω, ακολουθώντας μια προσέγγιση που είναι ευαίσθητη στον αφορά το φύλλο. Τι σημαίνει αυτό. Να μην εφαρμόζονται αυτές οι πολιτικές ουδέτερα. Δεν λέω ότι οι πολιτικές αυτές δεν μπορούν να έχουν θετική επιρροή ή αποτελέσματα σημαντικά για να αντιταχθούν στο φαινόμενο της ε, ανεργίας των νέων, που είναι ενδημικό φαινόμενο πλέον. Αλλά θα έπρεπε να αναλυθούν περισσότερο λαμβάνοντα υπόψη τη διαφορά με βάση το φύλλο. Δύο παραδείγματα. Πρόσφατε μελέτε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τη μαθητεία και τη χρήση της μαθητείας στην Ευρώπη έδειξαν το ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σχεδόν σε όλες τις χώρες στα διάφορα σχήματα μαθητείας που προωθούνται στα διάφορα κράτη-μέλη. Αυτό και πάμε στα προηγούμενα που αναφέρθηκαν λόγω διαχωρισμού με βάση το φύλλο. Διαχωρισμού με βάση την παιδεία. Χρησιμοποιούνται οι μαθητείες αυτές, τα προγράμματα μαθητείας σε τομείς που είναι περισσότερο αρσενική εντό εγωγικών από ότι φιλική. Δεν λέω ότι αυτό, με αυτό ότι δεν πρέπει να προωθούμε τη μαθητεία. Αλλά όταν προωθούνται πολιτικές που ευνοούν τη μαθητεία, θα πρέπει αυτές οι πολιτικές όμως να έχουν διαφορετικό αντίκτυπο. Θα πρέπει να εφαρμόζονται λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορά των φύλων. Ιδιαιτερότητες μεταξύ των δύο φύλων, διαφορών μεταξύ των φύλων. Και έτσι θα διαφοροποιηθεί και δυναμική και τα αποτελέσματα με βάση το φύλο. Παράλληλα, οι γυναίκες φαίνονται να εκπροσωπούνται καλύτερα σε άλλες φάσεις, πιο πολύ να είναι πιο σε άλλες προσπάθειες να εκπροσωπούνται καλύτερα. Αν δούμε καλύτερα τα δύο μέτρα, τις δύο διαδρομές που ακολουθούνται στον αφορά τη μαθητεία και την εκπαίδευση, με εξαιρέσει βέβαια που μπορεί να υπάρχουν στα διάφορα κράτη-μέρη, στις διάφορες νομοθεσίες. Λοιπόν, ε, ακολουθούνται διαδρομές που είναι λιγότερο προστατευμένες, οι ανεπίσημες μαθητής αν θέλετε, ε, ρυθμίζονται λιγότερα μέσω νομοθεσίας και κοινωνικής προστασίας. Ανεπίσημη μαθητή στο ΣΥΠΗΝ είναι αυτή. Και οι γυναίκες εκεί ε, εντάσσονται περισσότερο ε, και χρησιμοποιούνται αυτές οι ανεπίσημες μαθητείες ε, μέσω και πιο λιγότερο πιο συγκυριακής εργασίας Χρειάζεται λοιπόν καλύτερη προσέγγιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Χρειάζεται να προωθήσουμε μέσα από το πακέτο ε, ποιοτικό έλεγχο των διαφόρων ειδών μαθητείας. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη τη μεταβλητή του φίλου και εκεί, ούτως ώστε να καθορίσουμε καλύτερα αυτές τις προσεγγίσεις για να δούμε ποιες θα είναι οι διαφορετικές συνέπειες των διαφόρων δρομολογηθέντων μέτρων. Ένα άλλο παράδειγμα που μπορώ να αναφέρω είναι άλλες πολιτικές, όλα τα μέτρα της ενεργού πολιτικής εντός της αγοράς εργασίας που απευθύνονται προς τους νέους άντρες και γυναίκες, τους ανέργους και τους νετ άντρες και γυναίκες που δεν έχουν μπει στην αγορά εργασίας ούτε στην παιδεία που και σε αυτή την περίπτωση ε, έχουν διαφορετικά αποτελέσματα από αυτά που επιδιώκονται η ποικιλομορφία. σε πολλές αναλύσεις φαίνεται ότι χρησιμοποιούνται ε, με διαφορετικό τρόπο οι άντρες και οι γυναίκες μέσω διαφόρων τυπολογιών μέτρων. και έτσι υπάρχουν διαφορές και ιδιαιτερότητες όσον αφορά τις διάφορες παρεμβάσεις. Επ' αυτής της βάσης και με βάση αυτά τα παραδείγματα το σημείωμα που έχετε μιλούσαν πριν για μαθητείες και οικοτροφείο, χρήση οικοτροφείο για εκμάθηση. Ε, θα μπορείτε να βρείτε λοιπόν διάφορες λεπτομέρειες, διάφορους πίνακες που σας ενημερώνουν σχετικά με τα τρία πλαίσια που εθίγησαν και στις πρώτερες παρουσιάσεις δηλαδή την πτυχή που άπτεται της παιδείας, της μετάβασης από το σχολείο στη δουλειά και της ε, πτυχής που αφορά τη φροντίδα και την περίθαλψη. Όλα τα συμπεράσματα και οι συστάσεις που αναφέρονται σίγουρα υπογραμμίζουν, όπως προσπάθησα να επενθυμίσω στη δική μου παρουσίαση, το όφελος της χρήσης μιας προσέγγισης με βάση το φύλλο στις διάφορες πολιτικές και στην ανάλυση των φαινομένων. Σίγουρα στις λεπτομέρειες που αφορούν τις διάφορες συστάσεις θα βρείτε διαφορές πιο συγκεκριμένες, αλλά μπορούμε να εντοπίσουμε εκεί τρία μακροοφέλη σε μακροσκοπικό επίπεδο. Πρώτα απ' όλα, καλύτερη και πιο σωστή αντιμετώπιση και ανάλυση των στοιχείων και των φαινομένων. Χρησιμοποιώντας μια τέτοια προσέγγιση μπορούμε να προχωρήσουμε σε μεγαλύτερο βάθος, να καταλάβουμε καλύτερα τις δυναμικές που εμπεριέχονται σε κάποια στοιχεία και στην απλή παρουσίαση ενός φαινομένου και έτσι όχι μόνο για λόγους ισότητας αλλά για να έχουμε προστιθέμενη αξία δηλαδή θα καταφέρουμε μέσω της εμβάθυνσης να αντιληφθούμε καλύτερα τα φαινόμενα τα οποία έχουμε μπροστά μας και επί των οποίων θεσπίζουμε νομοθεσία και προγράμματα. Δεύτερον, κάτι πολύ σχετικό. Ε, χρειάζεται καλύτερη αντίληψη και κατανόηση των φαινομένων. Και έτσι μπορούμε να καταλήξουμε σε καλύτερο προγραμματισμό και μπορεί να ακολουθήσει μια καλύτερη εφαρμογή και των πολιτικών και των παρεμβάσεων. Και έτσι μπορούμε να απαντήσουμε στις πραγματικές ανάγκες, να καλύψουμε πραγματικές ανάγκες των νέων ανδρών και των νέων γυναικών. Τα παραδείγματα που προσπάθησα να συνοψίσω, αλλά όπως είδαμε και από όλες τις ομιλίες που προηγήθηκαν, είδαμε ότι ρίξαμε το φως στην προ στην οπτική γωνία του φίλου που μας επιτρέπει να δούμε πιο ξεκάθαρα πιο ακριβώς πώς μπορούμε να προγραμματίσουμε και να εφαρμόσουμε καλύτερα τις πολιτικές. Η παρέμβαση του νομοθέτη και η δρομολόγηση πολιτικών παρέμβασης που έχουν σαν σκοπό την αντιμετώπιση αναγκών που εκφράζονται από τον πληθυσμό Όλα αυτά πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι οι ανάγκες αυτές είναι διαφορετικές. Και πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ανάγκες των νέων γυναικών και των νέων ανδρών. Τρίτη μακροσκοπική θεώρηση των ωφελημάτων της σωστής προσεγγίσεως. Κάτι που συνδέεται με τα προηγούμενα άμεσα. Θέλουμε να καταφέρουμε. Α, έχω ένα άλλο λεπτό έτσι. Να μειώσουμε, να αμβλύνουμε τις αρνητικές συνέπειες, απροσδόκητες συνέπειες που θα μπορούσε να έχει μια ουδέτερη προσέγγιση, δηλαδή με προσέγγιση που δεν λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φίλου σαν μεταβλητή για την ερμηνεία και την ανάλυση του φαινομένου και της αντιμετώπισης. Μπορεί να φέρει σε δυσκερή θέση το μισό πληθυσμό. Όπω αν εφαρμόσουμε μια πολιτική, υποστηρίζουμε ισχυρά σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο κρατών μελών μια πολιτική ή μια παρέμβαση, αν δεν την αντισταθμίσουμε με τη συνιστόσα του φίλου, μπορεί αυτή να έχει απροσδόκητα αποτελέσματα διαφορετικά από τα αρχικώς επιδιωκόμενα. Αν δεν λάβουμε δηλαδή υπόψη διαφορές. Πέρασε ο χρόνος, θέλω να σταματήσω εδώ. Είμαι στη διάθεσή σας προφανώς για άλλες ε, αν θέλετε. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε πολύ. Πιστεύω πως πραγματικά εργαστήκατε πάρα πολύ σκληρά για να μπορέσετε να συνοψίσετε όλα αυτά που ακούσαμε σήμερα το απόγευμα και φυσικά πιστεύω πως ε, επίσης ε, αναφέρατε πολύ καλά επιχειρήματα όσον αφορά την ευαισθητοποιημένη προσέγγιση στην ανεργία των νέων. Σε όλα βέβαια χρειάζεται ευαισθητοποιημένη προσέγγιση θα έλεγα εγώ, αλλά ναι και σε αυτή. Τώρα θα γυρίσω στα ειδικά για να κάνω τα τελικά σχόλια προτού ολοκληρώσουμε αυτό εδώ το σεμινάριο. Εγώ θεωρώ ότι σήμερα το απόγευμα έγινε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ακούσαμε πολύ καλές ε, παρουσιάσεις ε, παιδαγωγικού χαρακτήρα. Εξετάσαμε το ζήτημα από πολύ διαφορετικές οπτικές γωνίες ε, είχαν παρουσιάσει σε πολλά και ενδιαφέροντα μέρη. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω και όλους όσοι συνέβαλαν στην ε, δική μας εργασία των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διότι χρειαζόμαστε άμεση επαφή και ενημέρωση σε σχέση με αυτά που προσπαθούμε να κάνουμε. Και ξέρετε, σας δείχνω εδώ ότι υπάρχουν περιλήψεις ε, των στοιχείων ε, που ναι. ακούσατε κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων και θα ήταν ίσως χρήσιμο να προμηθευτείτε αυτούς τους οδηγούς ε, για τις μελλοντικέ σας εργασίες. Υπάρχουν εδώ στην αίθουσα. Πέραν αυτού θα ήθελα να πω ότι ναι. είναι επιτακτική ανάγκη να ενισχύσουμε τη συνειδητοποίηση του ρόλου που παίζει η συνιστόσα των φύλων σε διάφορες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είδαμε πολλές στατιστικές, πολλά αριθμητικά στοιχεία και πιστεύω ότι ο συμπολογισμός αυτής της συνιστόσας, η προϋπόθεση, εκ των όνων κάνευ προϋπόθεση, είναι να ξεκαθαρίσουμε σε ποιους τομείς έχουν σημασία αυτές οι διαφορές και που δεν έχουμε στη διάθεσή μας τέτοια στοιχεία άρα θα πρέπει να τα προμηθευτούμε. Χρειαζόμαστε την ενσωμάτωση του παράγοντα φύλου σε όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, κατά την άποψή μου και είναι ιδιαίτερα αισθητή η ανάγκη του να υπάρξουν οι κατάλληλες κοινωνικές υποδομές τόσο ώστε να καταστεί δυνατή η αλλαγή του ρόλου των γυναικών, η μεγαλύτερη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας. Δυστυχώς σήμερα είναι καταδικασμένες στο να φροντίζουν παιδιά ή άλλα μέλη της οικογένειας λόγω της έλλειψης αυτών των υποδομών. Αυτό είναι ιδιαίτερα λυπηρό. Τέλος, και δεν θέλω να το ξεχάσουμε, ε, υπάρχουν και άλλα ζητήματα που σχετίζονται με αυτά τα κοινωνικά ζητήματα αλλά και με την ε, βαθύτερη οικονομική κρίση που είναι μία από τις αιτίες ε, του προβλήματος. Ακόμη και εάν κάναμε τα όλα όσα μας πρότειναν οι εμπειρογνώμονες, δεν σημαίνει ότι θα μπορούσαμε να επανορθώσουμε όλα αυτά τα προβλήματα, βαθύτερα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η κρίση. Με αυτό το καταληκτικό σχόλιο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές του πάνελ, όλους τους ακροατές. Γενικά ευχαριστεί και εμάς τους διερμηνείς ο Πρόεδρος, γιατί χάρη σε αυτού συνεχίζει μπορώ να μιλάω σου ειδικά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους ιδιαίτερο την Έρικα και το Policy Department του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διότι έκανε την πρακτική δουλειά, οργάνωσε και το πρόγραμμα της ακρόασης, συνέλεξε το υλικό. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για αυτή την μισή μερίδα μελέτης και στο επανειδήν.